Bueno, vamos a empezar. Buenos días Ας ε, ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, έχετε νομίζω μπροστά σας την ε, ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Περιμένουμε βεβαίως ακόμα την κυρία Βεζιά, αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε με κάποιες ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα. Θα ήθελα να εκφράσω εξ ονόματος της Επιτροπής την αλληλεγγύη μας ε, και τα συλληπιτήριά μας ε, για τα θύματα νεκρούς και τραυματίες ε, στον Ισημερινό. αρχίζει σιγά σιγά η διεθνής αλληλεγγύη να οργανώνεται, αλλά θα θέλαμε οπωσδήποτε και εμείς να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας με τον λαό του σημερινού. Αυτά για τα δυσάρεστα. Τα ευχάριστα. Όπως ξέρετε, χτες ο Αριφίτ και η Λεϊλά Γιουνούς ε, ελευθερώθηκαν δύο άτομα για τα οποία παλεύουμε εδώ στο Κοινοβούλιο σχεδόν δύο χρόνια τώρα. Και επιτέλους ε, απελευθερώθηκαν. Συνάντησαν ε, χτες και την κόρη τους, την ε, Ντινάιρα την οποία έχουμε γνωρίσει εμείς χρειάζονται βεβαίως και ιατρική φροντίδα αλλά τουλάχιστον είναι ελεύθερη και τώρα είναι σε καλά χέρια, στα χέρια των γιατρών. Λοιπόν, στην τελευταία Ολομέλεια στο Στρασβούργο το Κοινοβούλιο ενέκρινε τρία ψηφίσματα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Ένα για το Πακιστάν που αφορούσε ιδιαίτερα την επίθεση αυτή, την, την ε, επίθεση στην Ονδούρα και την κατάσταση των υπηρεσιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ξέρετε ότι το απόγευμα έχουμε και την ακρόαση για την αρπαγή γης και την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλών ανθρώπων ε, σε διάφορα μέρη της Ιφιλίου. Έχουμε βεβαίως, θα έχουμε και την κόρα της ε, κυρίας ε, Κασαρίς, η οποία έχει γίνει σύμβολο του αγώνα και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων για τη γη τους και θα έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί της κάποιες σκέψεις για την κατάσταση στην Ονδούρα η οποία οπωσδήποτε δεν έχει βελτιωθεί, να μην πω ότι έχει επιδεινωθεί κιόλα τελευταία. Επίσης το Κοινοβούλιο έκανε ένα ψήφισμα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος για την Ιγυρία και για άλλα ζητήματα που μας απασχολούν. Είχαμε τις εκθέσεις του 2015 για την Τουρκία, Αλβανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη μιας παγκόσμιας προσέγγισης για τη μετανάστευση και η έκθεση για την αναθεώρηση της στρατηγικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κεντρική Ασία. Λοιπόν, σήμερα το πρωί έχουμε το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Βερζιά για ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση στις τρίτες χώρες. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, κυρία Βεζιά για τη δουλειά που έκανε και να την ενθαρρύνω να συνεχίσει το έργο της γιατί νομίζω πως πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα και έχετε τον λόγο σας ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε για την καθυστέρηση κυρία Πρόεδρε υπάρχουν κάποια προβλήματα στην κίνηση δεν ξέρω αν ε, μιλήσατε για τα άσχημα νέα. Είχαμε το ναυάγιο αυτό στην ε, Μεσόγειο με 400 ε, νεκρούς. Καλό είναι να σκεφτούμε λίγο αυτούς τους ανθρώπους, άντρες, γυναίκες και παιδιά. Δεν είναι σίγουρο ακόμα το τι συνέβη. Ήταν κυρίως οι άνθρωποι αυτοί οι Σομαλοί και γενικότερα από το κέρας της Αφρικής και Σουδανοί. Θεωρώ λοιπόν πως η κατάσταση στις ε, χώρες αυτές, ε, είναι στο κέντρο της ε, έκθεσής μας ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδης ηγητές που είχα την ευκαιρία να συναντήσω και όλους μαζί και έναν έναν για το σύνολο των τροπολογιών έχουμε 300 τροπολογίες οπότε έχουμε δουλειά, δουλειά ακόμα μπροστά μας για να επιτύχουμε κάποια συνένεση. Ήδη έχω εξετάσει και συντάξει γύρω στις 20 συμβαστικές ε, τροπολογίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ε, γραμματεία και τους ε, συνεργάτες της ομάδας μου και τους δικούς μου τους βοηθούς Συνολικά θεωρώ πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποιον συμβιβασμό για τα περισσότερα από αυτά τα σημεία. Αν καταβάλουμε όλοι οι προσπάθειες, νομίζω εξάλλου ότι όλοι έχουμε συμφέρον να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερη συνένεση. Θα ήθελα απλά να επισημάνω κάποια σημεία. Όπως είπατε κυρία Πρόεδρε υπάρχει μια έκθεση η οποία εγκρίθηκε στην όλο μέλη για τη μεταναστευτική πολιτική της Ένωσης. Ε, στόχος δεν είναι να επαναλάβουμε λοιπόν τα όσα ήδη έχουν υποθεί, αλλά να επικεντρωθούμε στα προβλήματα της μετανάστευσης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες εκτός δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεδομένης της ε, παγκόσμιας κατάστασης μου φαίνεται πως αυτό το ζήτημα της μετανάστευσης ε, όπως ε, εξηγήθηκε ούτως ή άλλως ε, και στα εκτιμώντας είναι θέμα και ανθρωπινών δικαιωμάτων και εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης και μπορεί νομίζω να επηρεάσουμε, μπορούμε και εμείς να επηρεάσουμε θετικά τα ζητήματα αυτά. Κάποια προβλήματα που είχα ήδη επισημάνει στους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές ε, με κάποιες τροπολογίες οι οποίες αφορούσαν περισσότερο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι τις τρίτες χώρες. Και νομίζω ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Είμαι κάπως αισιόδοξη. Θα συναντηθούμε την επόμενη Τετάρτη για να κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για τις ε, συμβιβαστικές προτάσεις και να πω τέλος πως ε, θα ήθελα οι συμβαστικές προτάσεις ε, να συνταχθούν στα γαλλικά γιατί αυτή είναι η γλώσσα εργασίας μου. Δεν έχω ένα πρόβλημα να γίνουν μετά στα αγγλικά και γαλλικά, αλλά δεν μπορώ να εργαστώ στα αγγλικά, σε άλλη γλώσσα δηλαδή, πλην των γαλλικών, για να τα έχω τα πράγματα ξεκάθαρα στο κεφάλι μου. Μάλιστα. Θα δώσω τώρα τον λόγο στους ε, σκιώδεις ε, εισηγητές. Θα ήθελα να σας πω πως ε, δυστυχώς η επικεφαλής της γραμματείας εδώ πέρα μου λέει ότι είναι αδύνατον αυτό να γίνουν στα γαλλικά. Μα ε, κοιτάξτε, ε, είναι η γλώσσα της εργασίας μου. Δεν μπορώ να... Υποτίθεται ότι υπάρχουν 24 γλώσσες εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ελάχιστο είναι να σεβόμαστε τη γλώσσα των βουλευτών και τη εισηγητού. Ήδη έχω πρόβλημα με τις γλωσσικές διορθώσεις ε, στην αρχική μου έκθεση. Δηλαδή εκπλήσωμαι όταν διορθώνω τα γαλλικά μου. Ε, και υπάρχουν κάποια όρια στο θέμα το γλωσσικό εδώ μέσα. Δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε και ένα κείμενο στα αγγλικά. Εγώ θέλω να εργαστώ στο κείμενο το γαλλικό και θα ήθελα ή βασική έκδοση να είναι η γαλλική, γιατί εγώ δεν ξέρω να τα πω ακριβώς αυτά τα πράγματα και αν συμφωνώ ή διαφωνώ ή όχι, παρά μόνο στα γαλλικά. Ναι, ναι, βεβαίως. Ε, λέει η πρόεδρος, έχετε δίκιο. Και εγώ είμαι θύμα της επιβολής ε, των Αγγλικών στην δουλειά μας. Και όταν μου είπαν εμένα να αναλάβω αυτή τη δουλειά, δεν μου είπαν ότι θα μου επιβάλλουν τα αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, η γραμματεία μου είπε ότι δεν υπάρχει χρόνος να τα στείλουμε για μετάφραση. Γιατί η συνάντησή σας είναι την Τετάρτη. Σας λέω και εγώ είμαι θύμα της ίδιας κατάστασης. Εγώ θα δουλέψω στα γαλλικά, λέει η κυρία Βεζιά. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε, εγώ στα γαλλικά θα δουλέψω. Εντάξει, λέει η πρόεδρος. Ωραία. Θα δούμε. Τι θα κάνουμε. Είναι λυπηρό πράγματι και απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, Τέρεζα Κάτσερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά της πάνω στη συγκεκριμένη αναφορά. Πιστεύω ότι δεν ήταν ε, εύκολο έργο το να σύνταξει μια τέτοια αναφορά και όσον αφορά τις ε, τροπολογίες υπάρχουν κάποιες ε, τροπολογίες οι οποίες δεν επικεντρώνονται ε, στην σχέση με τρίτες χώρες και δεν επικεντρώνονται επαρκώς ε, στις βασικές αιτίες της μετανάστευσης όπως ε, το οποίο ήταν και ο σκοπός της συγκεκριμένης αναφοράς. Γι' αυτό το λόγο ναι θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση σχετικά με το πώς να συνεχίσουμε με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορώ να σχολιάσω ακόμα τις συμβιβαστικές αν όμως παρουσιαστεί η συγκεκριμένη έκθεση στα γαλλικά θα υπάρχουν κάποια ζητήματα διότι θα χρειαστώ τη βοήθεια κάποιου ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει ότι όσα γράφονται ε, είναι σύμφωνα με, τις, ε, με τα όσα έχουμε συμφωνήσει. Έχω κάνει επίσης ένα αίτημα για τη συνάντηση της επόμενης Τετάρτης ε, να λάβει χώρα σε διαφορετική ώρα η ε, πρόταση λοιπόν ήρθε εχθές ε, και έχουν προγραμματιστεί άλλες δραστηριότητες για εκείνη την ώρα. Όμως ε, νομίζω μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες και αδειμονώ να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους σκιώδης για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης έκθεσης. Ένα τελευταίο τώρα σχόλιο. Η συγκεκριμένη έκθεση ε, είχε κάποιες δυσκολίες ε, τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε προσπαθήσει να το κάνουμε αυτό λαμβάνοντας υπόψη μας ο στόχος της έκθεσης να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των αιτιών της ε, μετανάστευσης και τις σχέσεις που έχουμε με τις τρίτες χώρες ενώ επίσης θέλουμε να επικεντρωθούμε και στο πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα βασικά αίτια της μετανάστευσης. Καλό λοιπόν η έκθεση να διατηρήσει αυτό το στόχο ή δάλλως μπορεί να καταλήξουμε με μια ε, έκθεση που ε, θα δημιουργήσει αντιπαραθέσεις με άλλες επιτροπές και να επηρεάσει την τελική μας ψήφο πάνω σε αυτό. Όπως και να έχει, ανυπομονώ να συνεργαστώ με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις. Ευχαριστώ πολύ, η κυρία Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα πορτογαλικά. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ ε, την κυρία Βερζιά. Φυσικά ε, υπήρχε κάποια πίεση στο όλο θέμα ε, ε, ήταν όμως παρόλα αυτά ευχαριστώ για μένα να συνεργαστώ με τους υπόλοιπους. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες, κάποιες θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα Ε, εμείς λοιπόν συμφωνούμε ε, στο ζήτημα της, ε, των αιτιών της μετανάστευσης. Το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό και φυσικά είναι και το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πώς είναι η κατάσταση σε τρίτες χώρες. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε διότι γνωρίζουμε τα αίτια. Με χαροποίησε όμως το ότι υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν μεγάλες διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις ε, τροπολογίες και σίγουρα θα τα καταφέρουμε. Το σημαντικό είναι και νομίζω ότι σε αυτό θα επικεντρωθούμε ε, ότι ε, το θέμα είναι η σημασία, η βασική σημασία είναι να επικεντρωθούμε στην καταπολέμηση του της λαθρομετανάστευσης, την προστασία των παιδιών και των γυναικών. Είναι λοιπόν λογικό από τη δική μου οπτική και αυτό θα πρέπει να είναι και η λογική που θα διέπει αυτή την έκθεση, η, το θέμα δηλαδή της ένταξης, του συμβασμού των δικαιωμάτων των μεταναστών. Έλεγα λοιπόν ότι περιμένω τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα καλό τελικό κείμενο με τη συνεργασία όλων. Σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριος Δεμεσμέκερ δεν είναι εδώ. Οπότε δίνω το λόγο στην κυρία Μπεθέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για την τεράστια προσπάθεια και την πολύ καλή θέληση της κυρίας Βερζιά που βρίσκεται στην ε, βάση αυτής της ε, έκθεσης και για το γεγονός ότι αυτή η έκθεση θα συμπληρώσει και θα δημιουργήσει μια προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της ε, γενικής έκθεσης που ε, εγκρίναμε όσον αφορά τη μετανάστευση. Πρόκειται για μια έκθεση, όπως είπε και η κυρία Βερζιά, που, για την οποία έχουν κατατεθεί άπειρες τροπολογίες. Ελπίζω και ξέρω μάλλον πως θα είναι περίπλοκη η εργασία για την εξέφραση συμβαστικών λύσεων. Εγώ προσωπικά έχω υποβάλει διάφορες τροπολογίες, αλλά εμπιστεύομαι απόλυτα την κυρία Βερζιά ότι θα τα καταφέρει να φτάσει στο πνεύμα συνένεσης το οποίο θα πρέπει να καταλήξουμε με αυτή την έκθεση και ότι οι συμβαστικές τροπολογίες θα καταφέρουμε να ε, περιέχουν αυτή την προστιθέμενη αξία ε, που θα ε, τονίσουν αυτή, θα τονίσει αυτή την έκθεση. Εγώ από τη δική μου πλευρά θέλω να τονίσω κάποιες πτυχές για τις οποίες κατέθεσα τροπολογίες γιατί πρόκειται για πτυχές που πιστεύω ότι πρέπει να φωτιστούν περισσότερο. Από τη μια πλευρά ο βασικός στόχος ήταν να θεσπίσουμε και να μάλλον το νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των μεταναστών και να υποβάλουμε την γενική προβληματική ε, που αφορά αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο πιστεύω θα πρέπει να είναι σαφές, όπως είναι η αναφορά σε αυτούς τους ανθρώπους, να καταλάβουμε δηλαδή και ότι συμπεριλαμβάνονται εδώ όλοι οι άνθρωποι και να μην γίνεται συγκεκριμένη αναφορά μόνο σε ένα τμήμα αυτών. Έπειτα, Έχουμε προκλήσεις ε, όσον αφορά τους μετανάστες και αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ότι οι εθνικές κυβερνήσεις ε, και οι διάφορε, τα διάφορα κόμματα θα πρέπει να πάψουν να κατηγορούν ε, τους μετανάστες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ένταξη των μεταναστών και για την ανάπτυξη των χωρών μας. Επίσης θέλησα να συμπληρώσω κάποιες παραγράφους που αφορούν τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, ειδικά τα παιδιά και ως προς αυτό έχω καταθέσει τροπολογία όσον αφορά την ε, εμπορία ανθρώπων και ε, δηλαδή παιδιών και γυναικών κυρίως που είναι και τα βασικά θύματα. Πάντως γενικά πιστεύω πως ε, η ο άξονας της έκθεσης είναι σωστός ε, όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και θα ζητήσω από την κυρία Βέρζια να έχουμε όσο γίνεται πιο σύντομα τις συμβιβαστικές τροπολογίες ώστε να μπορέσουμε να τις μελετήσουμε και να τις εντάξουμε σε αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοράο δεν είναι εδώ, η κυρία Σαργεντίνη. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την κυρία Βέσια για την δουλειά που έχει κάνει μέχρι στιγμής ε, για το ότι προσπάθησε βεβαίως να συμβιβάσει τρεις-τέσσερις ε, τροπολογίες ε, σε μια συμβαστική τροπολογία που θα είναι ακόμα προοδευτική. Εμείς έχουμε καταθέσει κάποιες τροπολογίες οι οποίες αφορούν τα εμβάσματα γιατί αναγνωρίζουμε τον ρόλο των εμβασμάτων στις τρίτες χώρες και υπάρχουν οι δυσκολίες τελευταία ε, στο πρίσμα της χρημα... στο, πλαίσιο, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της ε, τρομοκρατίας όσον αφορά την αποστολή εμπασμάτων ειδικά για όσους προέρχονται και κατάγονται από τη Σομαλία και δύσκολα μπορεί να στείλει κανείς λεφτά στη Σομαλία τα δικαιώματα επίσης ε, των οικονομικών μεταναστών ε, και τα δικαιώματα τους στις χώρες, προστασία τους στην κοινωνία που τους φιλοξενεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν λιγότερα δικαιώματα κατά την άποψή μου. Το θέμα των πολλών υπηκοτήτων, ε, πολλοί, περισσότεροι άνθρωποι πλέον έχουν πάνω από ένα διαβατήρια και βλέπουμε σε μια συζήτηση που γίνεται πιο εθνικιστική πως οι χώρες προσπαθούν να αγνοήσουν ένα από τα διαβατήρια ή μάλιστα να να απαγορεύσουν ε, την δεύτερη υπηκότητα, κατά οποίο είναι αδύνατον όταν βλέπουμε ε, πως οι οικογένειες γίνονται όλο και πιο ε, πολυεθνικές. Το θέμα των απάτριδων, η πατερμοστία του η ξεκίνησε μια εκστρατεία, το θέμα των εσωτερικά εκτοπισμένων, που επισήμως δεν είναι μετανάστες, αλλά έχουν καταφύγει στη δική τους χώρα, κάπου αλλού, που συχνά το παραμελούμε. Η κράτηση μόνο και μόνο γιατί κάποιος είναι μετανάστης ε, και ειδικά η κράτηση ανηλίκων είναι πράγματι ε, ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε τρίτες χώρες αλλά και εμείς κρατούμε παιδιά εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παρακολούθηση των επιστροφών από την Ευρώπη σε τρίτες χώρες, η εκτός της Ένωσης πώς θα διασφαλίσουμε τη σωστή υποδοχή τους ε, με ανθρώπινα δικαιώματα και τέλος τα δικαιώματα όσων ε, δεν έχουν έγγραφα σε μια κοινωνία, που, ε, κατά το οποίο οδηγεί σε τεράστια σκάνδαλα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, ξέρω πως έτσι ο κατάλογος σας γίνεται μακρός και ελεύθερος, αλλά θα ήθελα να βρούμε κάποιες λύσεις στις ε, συμβαστικές σας Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σαρτσεντίνη. Τώρα θα δώσω το λόγο στον υπεύθυνο, στην υπεύθυνη μάλλον της Επιτροπής Ανάπτυξης για αυτή την έκθεση, ε, η κυρία Αλμπιόλ. Ε, Καταρχά να ευχαριστήσω την Κριστίνη Βεριζιά και ολόκληρη την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη δουλειά που κάνετε με αυτή την έκθεση και από την Επιτροπή ΔΕΒΕ, της ανάπτυξη δηλαδή, προετοιμάζουμε μια γνωμοδότηση για να σας ε, δώσουμε ποια είναι η άποψη αυτή τη επιτροπή μα. Καταρχά, τονίζουμε ότι η αναγκαστική μετανάστευση, δηλαδή ο κόσμο που αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του για οικονομικού ε, πολιτικού ή κοινωνικούς λόγους, είναι ε, θέμα το οποίο επιβαρύνει από άποψη ευθύνη τη Κομισιόν, γιατί πολλέ φορέ όλα αυτά τα προβλήματα οφείλονται στι δραστηριότητε των πολυεθνικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στι εμπορικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση στι τρίτε χώρε, που οδηγούν ε, στην ε, φτώχεια του πληθυσμού και την, αδε... την... στην εκμετάλλευση, εκμετάλλευση των πόρων των χωρών αυτών. Επίση, τονίζουμε ότι πολλά κρατημέλη παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα σε αυτέ τι ξένε χώρε, στι χώρες μάλλον αυτές ε, της μετανάστευσης και τονίζουμε και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ε, ακριβώς ε, έχει παροτρύνει τη χρέωση χωρών ε, το εξωτερικό χρέος των χωρών αυτών αυξάνεται και λόγω των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι χώρες πια αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους. Έχουμε, ε, μιλάμε επίσης για τα κέντρα κράτησης, για τους μετανάστες και πως αυτοί πέφτουν θύματα απελάσεων, ε, νομικών παραβιάσεων, παραβίασης των δικαιωμάτων τους για την υγεία και την παιδεία. Επίσης κάτι ακόμα πολύ σημαντικό που θέλουμε να σας διαβιβάσουμε από την Επιτροπή Ανάπτυξη είναι ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταμεία ανάπτυξη για να το, ε, χρηματοδοτηθούν πολιτικέ μετανάστευση. Πολλέ φορέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν χρησιμοποιηθεί αναπτυξιακά κονδύλια στην ουσία για να επιβληθούν σε τρίτε χώρε μεταναστευτικέ, εμπορικέ, οικονομικέ πολιτικέ. Και επίση τέλο ε, αυτό που θέλουμε και διζητάμε είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακαλέσει και μάλιστα επιγόντω κάθε είδο συμφωνία μεταναστευτική με τρίτε χώρε των οποίων οι χώρε παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω πω αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σε αυτή την κατάσταση εφόσον έχουμε υπογράψει και ε, υπογράφηκε και αυτή η συμφωνία της ντροπή μεταξύ Ένωσης και Τουρκίας. Ε, οι τροπολογίες έχουν ήδη κατατεθεί, οι συμβιβαστικές έχουν επίση κατατεθεί στη δική μα Επιτροπή και απόψε θα ψηφίσουμε για τι τροπολογίε στην Επιτροπή ανάπτυξη και για την γνωμοδότηση και θα σας διαβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αλβιόλ. Ο κύριος Πανζέρη ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγγνώμη δεν άκουσα την εισήγηση της Μαρή Κριστίν. Απλά θέλω σε αυτή τη σημαντική έκθεση να μην είμαστε εκτός τόπου σε σχέση με την συζήτηση που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προχτές μόλις στο Λουξεμβούργο οι Υπουργοί Εξωτερικών συνεδρίασαν. Υπάρχει μια πρόταση ε, και θα ήταν σκόπιμο να ενταχθεί σε αυτήν την, την έκθεση σε σχέση με το Σύμφωνο Μετανάστευσης ε, Migration Compact. Ε, δηλαδή πρόκειται για μέσα χρηματοοικονομικά τα οποία θα απευθυνθούν στις τρίτες χώρες ακριβώς ώστε να αποφευχθεί η η αύξηση της μεταναστευτικής ροής σε βαθμό ώστε να μην μπορούμε πια να την αντιμετωπίσουμε. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποια παραπομπή σε αυτήν τη συζήτηση μέσα στην έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά έχει να σχολιάσει κάτι. Εγώ νομίζω πως... δεν κατάλαβα καθόλου τι μου ζήτησε ο κύριος Παντζέρη. Παντζέρη δηλαδή. Ε θα τα πούμε μεταξύ μας για να συνοηθούμε. Ευχαριστώ το, όλους τους σκιώδεις. Τα όσα άκουσα μάλλον επιβεβαιώνουν αυτή μου την ιδέα ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Πάντως, ε, εγώ θέλω να υποβάλω όσο γίνεται περισσότερες συμβιβαστικές, ώστε ακριβώς ε, να ε, συμπεριλάβω τις απόψεις όλων. Όπως σας είπα, Ήδη έχω περίπου προετοιμάσει μάλλον μου προτίμασαν και εγώ επικυρώνω, επικυρώνω τώρα καμιά εικοσαριά τροπολογίες και ε, μέλημά μου είναι να προσπαθήσω να συγκεντρώσω όσο γίνεται περισσότερες. Γιατί όσο περισσότερες τροπολογίες έχουμε εκτός συμβιβαστικών, τόσο περισσότερη απογοήτευση θα έχουμε ε, από όλους. Βεβαίως, το σημαντικό θέμα είναι η προστασία των μεταναστών και των δικαιωμάτων τους. Αυτό είναι μόνο ένα στοιχείο όσον βέβαια σε σχέση με τις βαθύτερα, τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, διότι οι μεταναστευτικές ροές έχουν διάφορα και ποικίλα αίτια. Δεν πρέπει να ε, παγιδευτούμε στη συζήτηση μετανάστες, ίσως ε, η οικονομική μετανάστευση πρόσφυγες. Στις περισσότερες χώρες ε, το δικαίωμα στο άσυλο δεν υπάρχει. Η εφαρμογή της σύμβασης της, μάλλον η σύμβαση της Γενέβης δεν είναι καν υπογεγραμμένη και όταν υπογεγραμμένη δεν μεταφράζεται σε πράξεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να υπάρξουν νομοθεσίες που προστατεύουν τους μετανάστες και που επιτρέπουν το δικαίωμα ασύλου. Πρέπει πραγματικά να προσπαθήσουμε και μονίμως να προσπαθούμε να ε, μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων στις τρίτε χώρες και να μην τα βλέπουμε όλα με τα δικά μας, από τη δική μας μονοπτική γωνιά. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν ακούγονται προς τα έξω. Θα πρέπει καταρχάς λοιπόν να τα συζητήσουμε με τις έξω κυβερνήσεις αλλά και με όσους ασχολούνται με αυτά τα θέματα εκεί. Τώρα ξέρω ότι έχουμε συζήτηση με την κυρία Μπεσέρα όσον αφορά την ε, χώρα των μεταναστών. Για μένα ε, μάλλον, το θέμα των απάτριδων είναι ένα θέμα για τη μετανάστευση και η συνέπεια της μετανάστευσης. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν εθνικότητα διότι δεν έχουν ε, νομικό καθεστώς στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Άρα λοιπόν και εδώ πρέπει να βρούμε μια συμβιβαστική η οποία να μην σημαίνει κατάργηση κάθε αναφορά στους απάτες γιατί κάτι τέτοιο δεν θα ικανοποιεί την ε, παρακαθήμενή μου η οποία έχει υποβάλει ένα σωρό τροπολογίες για αυτό το θέμα. Για, τώρα, για τις ε, ευάλωτες ομάδες ε, έχουν κατατεθεί ένα σωρό τροπολογίες και για τις γυναίκες και για τα παιδιά και φυσικά εδώ θα κάνουμε συμβιβαστικές δεν νομίζω πως θα έχουμε πρόβλημα να βρούμε κάποια συμφωνία. Και για το θέμα, τα θέματα κράτησης, η κράτηση θα πρέπει να είναι η εξαίρεση για τους μετανάστες και ακόμα περισσότερο για τους πρόσφυγες και ακόμα περισσότερο για τα παιδιά. Ε, οπότε και εδώ θα πρέπει να βρούμε μια κάποια διατύπωση ε, ώστε να σας καθησυχάσω. Υπάρχουν ε, ε, τροπολογίες, θα σας τις στείλω όσο γίνεται πιο σύντομα και στα γαλλικά και στα αγγλικά. Και το είπα και το Ξαναλέω ότι η γαλλική εκδοχή θα είναι η βασική. Το έχω πει και ξαναπεί ότι αρνούμε να εργαστώ στα αγγλικά. Έχω το αγγλικό κείμενο, την αγγλική εκδοχή, αλλά εγώ δεν είμαι βεβαία για το ότι εννοώ αυτό που λέω όταν είναι στα αγγλικά. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να θεωρηθεί βάση η γαλλική εκδοχή, ακόμα και αν μπορούμε να δουλέψουμε και στις δύο γλώσσες. Γιατί διαφορετικά θα κάνω και τροπολογίε γλωσσικέ που δεν θα σας ικανοποιούν και θα τσακώναμε με την γλωσσική υπηρεσία. Να σας διηγηθώ δύο, πρα... δύο ιστορίες τώρα. Τον Μάρτιο υιοθετήσαμε για το θέμα του φύλου και της ισότητας ανδρών και γυναικών στο, ε, ε, εντός στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο. επέμεινα ότι θα πρέπει το θηλυκό να γράφεται με ένα ε στο τέλος όπως είναι στο σωστό στα γαλλικά. Χρειάστηκε να τσακωθώ 100 φορές όταν είμαστε φεμινιστές στα γαλλικά η συγγήτρια, ραπορτέρ, γράφεται με ένα έ στο τέλος. Ακόμα και αν δεν είστε φεμινίστρια, γράφετε με ε. Στο τέλο. Εν πάση περιπτώσει, εξαρτάται τι σημαίνει φεμινίστρια. Α μην αρχίσουμε τέτοια συζήτηση τώρα. Πάντω, στα γαλλικά ε, γράφεται με ένα ε στο τέλο, ε, όταν είναι η συγγήτρια γυναίκα. Και επειδή είμαι γυναίκα, επέμεινα γι' αυτό και τσακώθηκα με τι γλωσσικέ υπηρεσίε 100 φορέ μέχρι να το δεχτούν. Τώρα, άλλο, άλλη ιστορία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο αγώνας που κάνουμε στα θέματα των δικαιωμάτων είναι, και τα γαλλικά είναι μια πολύ σεξιστική γλώσσα, δικαιώματα λέμε του ανδρός στην ουσία, ενώ είναι του ανθρώπου, Θέλουμε όταν λέμε droit de να γράφεται με κεφαλαίο άστο η λέξη όμα ώστε να διακρίνεται η λέξη άνθρωπος που σημαίνει και άνθρωπος από την λέξη άνδρας. Είναι ένα προβληματάκι αυτό γιατί αυτό αλλάζει τη φύση της σκέψης μου όταν εγώ δεν πάω καλά ή είναι οι γλωσσικές υπηρεσίες οι οποίες δεν καταλαβαίνουν τους λέω. Αυτό δεν έχει λυθεί το θέμα. Ε. Όχι, όχι ακόμα. Δεν ξέρω. Εγώ θα κάνω όσε τροπολογίε χρειάζεται για να επιβληθεί αυτό. Εγώ θέλω στα γαλλικά που εγώ συντάσσω στο κείμενό μου να γίνεται σεβαστή η γλώσσα μου και ο τρόπο με τον οποίο βλέπω τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό είναι και το φυσιολογικό. Ναι, είναι φυσιολογικό. Προχωράμε και ευχαριστώ και πάλι όλου και πιστεύω ότι το αργότερο αύριο ή την Παρασκευή θα έχετε μια πρώτη εκδοχή των συμβιβαστικών τροπολογιών, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να δουλέψετε. Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν η ψηφοφορία θα γίνει 23-24 στην ΑΦΕ. Δεν έχει αποφασιστεί. 23-24. Κύριε Χόουιτ, ξέρω ότι είστε πολύ γρήγορος. Ελπίζω να το αποδείξετε γιατί από, άποψη χρόνου τα πάμε χάλια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, όσο ε, πρώτος ο ε, ε, που έχει μητρικά, μητρική τα αγγλικά δεν νομίζω ότι πρέπει να επιβάλλεται η γλώσσα αυτή σε όλους και ε, χαίρομαι για το γεγονός ότι μιλάμε ε, για το φεμινισμό ε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υποστηρίζεται στις εκθέσεις μας ε, ασχέτως του πώς γράφεται η λέξη συγητή ή συγγήτρια. Ας μιλήσουμε τώρα ε, για, το, για την έκθεση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Θα ήθελα να πω ότι η Στίβενς κάνει πάρα πολύ καλή ε, δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Οι υπόλοιποι γνωμοδότες συνεισέφεραν ε, πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ καλά στο θέμα αυτό. Σε όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες τις οποίες έχω παρουσιάσει, όπως εξήγησα στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων, επίτηδες δεν ε, αναφέρθηκα σε κάποια γλωσσικά ζητήματα και αυτό αφορά τις τροπολογίες 1, 6, 16, 15 και 20. Αυτά αφορούν τις ανθρωπιστικές καταστροφές, όμως ορισμένοι συνάδελφοι έχουν σχόλια για αυτό ε, σχετικά με τα δεδομένα και κάποιοι συνάδελφοι έφεραν τροπολογίες πάνω σε αυτά. Θα ε, κάνω ε, συμβιβαστικές πάνω σε αυτά για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες αυτές τις ε, περιοχές. Τώρα όσον αφορά τους συνάδελφους από το EPP, με τον συνάδελφο Κώσα υποστηρίζω τις τροπολογίες τους και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ποιο είναι το σωστό σημείο για τις συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις όλα αυτά συνδύονται σχετικά με την μη χρηματοδότηση ε, ζητημάτων ε, παρά τη χρηματοδότηση και νομίζω ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποια σύγχυση. Ε, στο 21 υποστηρίζω τα δεδομένα και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν ο κυρία Ντεσμάκερ τώρα η ε, τροπολογία 4 σχετικά με την, ε, με την ε, επικουρικότητα είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να συμπεριληφθεί. Για την 8 τώρα θα πρέπει να συμπεριληφθεί και τη 13 υποστηρίζω και θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη συμβιβαστική μαζί με την 14 της κυρίας Βαλένσια στη 15 σχετικά με την πρόσβαση και την προσβασιμότητα. Την υποστηρίζω, όμως ε, θα πρέπει να έχουμε και μια συμβιβαστική με αυτές ε, για τη 18 για το οικογενειακό περιβάλλον, αντιλαμβάνομαι το νόημα. Τώρα αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί, δεν ξέρω αν ταιριάζει με τη συγκεκριμένη έκθεση, θα πρέπει να το συζητήσουμε. Και 26 το θέμα είναι καθαρά γλωσσικό και υποστηρίζω το θέμα. Ο κύριος Κράουν και πάλι ε, για την 3, 5 και την 28 υποστηρίζω το θέμα. Την 9 σχετικά με τη χρηματοδότηση θα συμπεριληφθεί στη συμβαστική και 28 θα υπάρξει μια ε, προσθήκη. Ο κύριος Κοπτσέφ σχετικά με την τροπολογία 10 για τα διαρθρωτικά ταμεία. Μου άρεσαν κάποιες από τις ε, τροπολογίες θα συζητήσουμε για αυτό και η 29 με την ανάπτυξη την υποστηρίζω όμως υπάρχει μια άποψη της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης που θα πρέπει να, να την συζητήσουμε και τώρα όσον αφορά τα ζητήματα φεμινισμού και δικαιώματα γυναικών η κυρία Βαλένσια ε, παρουσίασε μια πάρα πολύ καλή τροπολογία σχετικά με την προσφασιμότητα την υποστηρίζω, είναι πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να υπάρχει μια συμβαστική με αυτά τα δύο. Αυτή ήταν η προσίασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χόουιτ, ο κύριος Τζιμ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ ε, τον συναδελφό μου, κύριο Κοπάτσεφ, που δεν είναι εδώ και σας ευχαριστώ εκ μέρους του για το κείμενο της συγκεκριμένης έκθεσης. Συμφωνούμε ότι είναι ένα πολύ ισορροπημένο κείμενο, όμως δεν έχουμε τροπολογίες με τις οποίες ε, ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, περαιτέρω συζήτηση με τον εισηγητή και τους κοιόδες. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να τονίσουμε είναι το το ζήτημα μιας θετικής ε, γλωσσικής έκφρασης σε κάποια σημεία του κειμένου. Ο ίδιος ε, το τόνισε αυτό. Να υπάρχει δηλαδή ένα πιο θετικό λεξιλόγιο το οποίο να μπορούμε να αποδεχθούμε το ζήτημα των διαρθρωτικών ταμείων τώρα και η χρήση αυτών το συζητήσαμε και αυτό θέλουμε να τονίσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δωρητής ε, της αναπτυξιακής βοήθειας και θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο έγγραφο θα πρέπει να αναφερόμαστε στις πολυμερείς σχέσεις ε, και θα πρέπει να το τονίσουμε. Υπάρχει αυτή η χρηματοδοτική ε, προσπάθεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη. Αυτά λοιπόν πιστεύω ότι είναι τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία αναφέρει ο κ. Κοβάτσεφ, τα οποία παρουσίασα εγώ με βάση το έγγραφο που μας έστειλε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Πασταβίτσιους. Αρχικά, ο Σκιώδης δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σήμερα. Το κείμενο του κυρίου ε, Χόβιτ. Θα μιλήσω λοιπόν ε, εκ μέρους του ε, παρόλο ε, που είναι έμπειρο μέλος του Κοινοβουλίου. Ο κ. Ρίτσαρτ δεν μπόρεσε να παρουσιάσει κάποιες τροπολογίες, σεβόμενος πάντα την πολύ καλή δουλειά που κάνατε. Βλέπουμε την, το έγγραφό σας ως πολύ ισορροπημένο. Θα το εξετάσουμε και θα λάβουμε υπόψη μας τις τροπολογίες που αναφέρετε. Καλή σας επιτυχία. Είναι ένα πολύ έγγραφο πάνω στο, οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε και επίσης είναι ένα καλό παράδειγμα, ε, διότι η αγγλική γλώσσα μπορεί να είναι μια γλώσσα πάνω στην οποία μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε συμφωνίες. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Χάουιτ, έχετε κάποιο τελικό σχόλιο? την ε, γλώσσα σας. Εγώ για να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο θα, ήθελα να πω ότι και δύο εκθέσεις τόσο της κυρίας Βεριζιά όσο και του κυρίου Χάουιτ είναι εκθέσεις που έχουν γίνει ε, ενδελεχώς έχουν εμβαθύνει και στα θέματα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε. Ελπίζω πως θα φτάσουμε όντως σε ευρύες ε, συνενέσεις ώστε να έχουμε ε, στήριξη και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συγχαίρω τους δύο εισηγητές. Thank you very much και merci beaucoup. Γεια σας κύριε Χόβιτ. <laughs> Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας μας διάταξης που είναι σημαντικό. Είχαμε προβλέψει ανταλλαγή απόψεων με την ε, κυρία που με συνοδεύει στα αριστερά μου, την κυρία Τασλίμα Νασρίν, που είναι συγγραφέας από τον Μπαγκλαντές και τιμήθηκε με το βραβείο Σαχάροφ το 1994. Δεν είναι εύκολο να κάνουμε σύντομη παρουσίαση της κυρίας Νασρίν γιατί είναι μια ιστορική αγωνίστρια κατά της ε, θρησκευτικής ακρότητας αλλά και κατά της ε, καταπίεσης των γυναικών. Έχαμε κι άλλον έναν ε, καλεσμένο, τον κύριο Σαλή Οσμάνα που δεν μπόρεσε να ταξιδέψει γιατί οι αρχές του Σουδάν ε, του έχουν ε, αφαιρέσει το διαβατήριο. Έπρεπε να ταξιδέψει στη Γενέβη καταρχάς και μετά δεν μπόρεσε Δεν μπορέσαμε να του στείλουμε γρήγορα θεώρηση και έτσι δεν μπόρεσε να έρθει. Ο κύριος Σωσμάν έχει στείλει μια ανακοίνωση, αλλά δεν την έχω την ανακοίνωση αυτή. Όταν θα την λάβω θα σας την διαβιβάσω. Θα δώσουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Νασρίν που είναι εδώ στο πλαίσιο του φεστιβάλ κινηματογράφου One World. Είναι μέρος των ειδικών που συζήτησαν τη φιλμ Μάγι του που αναφέρεται στις 19 Απριλίου που αναφέρεται στην ριζοσπαστικοποίηση ειδικά στο Βέλγιο. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Νασρίν που ήρθατε και θα σας ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανησυχώ πάρα πολύ για τον Μπαγκλαντές και την Ινδία. Ξέρετε τι συμβαίνει. Ο Ισλαμικός ε, φονταμεταλισμός προχωράει, οι φονταμεταλιστές προ, σκοτώνουν ε, ανθρώπους οι οποίοι είναι υπέρ του κοσμικού κράτους, οι οποίοι σκέφτονται ελεύθερα, μπλόγγερ, συγγραφείς, έχουν σκοτώσει ήδη πάνω από δέκα ταλαντούχους συγγραφείς και μπλόγγερ αλλά η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές ε, δεν ανέλαβε καμία δράση κατά των δολοφόνων δεν έκανε καμία ενέργεια Πιθανότατα θέλει η κυβέρνηση του να χρησιμοποιήσει την θρησκεία για τα δικά της ε, συμφέροντα. Πιθανότατα ο Πρωθυπουργός Εικασίν θεωρεί ότι Πρωθυπουργός με θεωρεί ότι αν ζητήσει από την αστυνομία να συλλάβει τους δολοφόνους θα χάσει ε, ψήφους από τις ε, θρησκευόμενες ε, μάζες. Οπότε δεν υπάρχει δικαιοσύνη για τους διαφωτισμένους αυτούς blogger και συγγραφείς. Ανταυτού η Πρωθυπουργό λέει ότι κανείς δεν θα πρέπει να θίγει το θρησκευτικό αίσθημα των πολιτών. Είναι όμως αναγκαίο στη χώρα αυτή να ασκήσουμε κριτική στις δογματικές πρακτικές της θρησκείας. Οι γυναίκες υποφέρουν υπό το Ισλάμ. Έχουμε θρησκευτικούς νόμους οι οποίοι δεν ε, επιτρέπουν την ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Οι σε δεν έχουν ίσα δικαιώματα στο γάμο, το διαζύγιο, την επιμέλεια των παιδιών και την κληρονομιά γιατί έχουμε νομοθεσία η οποία βασίζεται στην θρησκεία, όχι στην ισότητα. Εμείς λοιπόν οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προσπαθούμε να αποκτήσουμε έναν αστικό κώδικα ο οποίος θα βασίζεται στην ισότητα αλλά βεβαίως η κυβέρνηση δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον για να μεταρρυθμίσει το Ισλάμ ή να επιφέρει κάποια αλλαγή. Οπότε δεν υπάρχει ελευθερία έκφρασης επίσης στο Μπαγκλατές γιατί βλέπετε ε, πως δολοφονούνται όσοι σκέφτονται ελεύθερα γιατί άσκησαν κριτική στο Ισλάμ και μόνο. Αν ασκεί κανείς κριτική σε άλλες θρησκείες δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά όποτε κάποιος ασκήσει κριτική στο Ισλάμ φυλακίζεται ή αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα όπως έκανα εγώ πριν από 22 χρόνια. Αναγκάστηκα να φύγω από τη χώρα μου γιατί οι φονταμεταλιστές δεν ήθελαν να ζήσω στη χώρα μου και η κυβέρνηση αντί να δράση κατά αυτών που εξέδωσαν φετφάδες εναντίον μου και με επικήρυξαν και όλες κινήθηκε εναντίον μου. Με κατηγόρησαν ότι έφυξα το θρησκευτικό αίσθημα και αναγκάστηκα να κρυφτώ γιατί με αναζητούσαν για να με συλλάβουν και τελικά ε, εκδιώχθηκα από τη χώρα μου. Πέρασαν 22 χρόνια. Δεν έχω δικαίωμα να επιστρέψω στη χώρα μου. Το πότε τώρα... μουσουλμάνοι φονταμεταλιστές ε, διαπράττουν φρικτά εγκλήματα. Θα με είχαν σφάξει κυριολεκτικά στο Μπαγκλαντές όπως και άλλους ε, συγγραφείς ε, που είναι υπέρ ε, του κοσμικού κράτους. Κάποιοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα, κάποιοι παραμένουν. Και δολοφονούνται. Και η κυβέρνηση αντί να κάνει κάτι για να κυνηγήσει τους δολοφόνους κυνηγά αυτούς τους blogger και τους διανοούμενους οι οποίοι ζητούν προστασία από την αστυνομία η οποία δεν τους δίνεται και μάλιστα τώρα κρύβονται κάποιοι από αυτού γιατί δεν είναι εύκολο να φύγει κανεί από τη χώρα γιατί δεν είναι εύκολο να πάρει βίζα για την Ευρώπη, την Αμερική ή τις γειτονικέ χώρες. Οπότε δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Ίσως ε, θα έπρεπε να πείτε στην Πρωθυπουργό του Μαγκλαντές να, να λάβει δράση κατά αυτών των ε, Ισλαμιστών δολοφόνων. Γιατί ξέρετε, πριν από 15 μέρες ένας άνθρωπος επειδή ε, ήταν υπέρ της λογικής και της εκοσμίκευσης δολοφονήθηκε από τους Ισλαμιστές. Γιατί σκοτώνουν τους ανθρώπους, γιατί ξέρουν ότι δεν θα συλληφθούν, δεν θα τους συμβεί τίποτα. Οπότε δεν φοβούνται και τίποτα. Οπότε τι θέλουν. Θέλουν να μην υπάρχει ελευθερία έκφρασης ε, για τους αντιπάλους τους. Δεν θέλουν να ακούσουν καμία κριτική του Ισλάμ, αλλά χωρίς κριτική στο Ισλάμ είναι αδύνατον να υπάρξει αλλαγή σε μια Ισλαμική κοινωνία. Ε, δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός ε, θρησκείας και κράτους που είναι κάτι το οποίο απαιτείται στις μουσουλμανικές χώρες. Ξέρετε κάποτε στις χριστιανικές χώρες οι χριστιανοί φονταμεταλιστές σκότωναν ε, όσους ε, ασκούσαν κριτική στο χριστιανισμό αλλά εσείς ε, διαχωρίσατε την εκκλησία από το κράτος υπήρχε μια αλλαγή αυτό δεν έχει γίνει στις Ισλαμικές χώρες οι γυναίκες υποφέρουν πολύ λόγω του Ισλαμικού δικαίου και των κανόνων. Στο Μαγκλαντές οι περισσότερες γυναίκες τώρα φοράνε μπουρκα και μαντήλες γιατί έχει ξεκινήσει ένας ε, μια ε, Ισλαμοποίηση και η κυβέρνηση δεν ε, κάνει τίποτα. Οι φονταμεταλιστές λαμβάνουν κονδύλια από τη Μέση Ανατολή, από Ισλαμιστές εκεί. Οπότε χώρα λοιπόν καταστρέφεται και όσοι είναι υπέρ μιας κοσμικής κοινωνίας ε, υφίστανται επιθέσεις και από τους Ισλαμιστές ε, και από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αντί να συλλάβει τους δολοφόνους, τους φονταμεταλιστές που εκδίδουν φετφάδες ε, κατά συγγραφέων που δολοφονούν ε, τους blogger κτλ. Συλλαμβάνει άθεους ε, και λογικοκράτες ε, και λοιπούς γιατί ασκούν κριτική κατά του Ισλάμ με τον νόμο περί βλασφημίας που υπάρχει και στην Ινδία και στο Πακιστάν. Οι νόμοι αυτοί περί βλασφημίας χρησιμοποιούνται από τα κράτη για να συλλάβουν όσους σκέφτονται ελεύθερα. Είναι λοιπόν μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, όχι μόνο στον Παγκλαντές, και στην Ινδία. Ίσως γνωρίζετε ότι οι Ινδουιστές φονταμεταλιστές πρόσφατα σκότωσαν κάποιους αθώους μουσουλμάνους γιατί έφαγαν μοσχάρι. Ή γιατί εμπορεύονται αγελάδες. και οι Ινδουιστές, οι φανατικοί, τους κατηγόρησαν ε, ότι έτρωγαν ε, το μοσχάρι και τους ε, κατέσφαξαν. Επειδή έτρωγαν μοσχαρίσιο κρέας και σκότωσαν και κάποιους οι οποίοι ήταν υπέρ της λογικοκρατίας επειδή άσχησαν κριτική στον Ινδουισμό. Και το λυπηρό είναι ότι η... Βεβαίω η κυβέρνηση της Ινδίας δεν έκανε τίποτα. Θεωρώ λοιπόν πως ε, και στην Ινδία ε, χρησιμοποιεί και εκεί πέρα η κυβέρνηση το, την ε, εκεί θρησκεία για τους σκοπούς της και επειδή δεν γίνεται τίποτα ε, κατά αυτών των δολοφόνων, των Ινδουιστών σε αυτή την ε, περίπτωση θα ρίνονται προφανώς για να διαπράττουν αυτά τα φρικτά εγκλήματα. Οπότε δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εγώ συγγραφέας είμαι. Γράφω κατά του εξτρεμισμού, κάθε είδους ε, και του φανατισμού. Και είμαι υπέρ ενός ενιαίου αστικού κώδικα που δεν θα βασίζεται στη θρησκεία για να μην υποφέρουν οι γυναίκες από τους θρησκευτικού νόμους. Είμαι υπέρ της ε, κοσμικής ε, εκπαίδευσης ε, και όχι της θρησκευτική. Ίσως ξέρετε πως τα τζαμιάκι με ντρεσέδες στον Μπαγκλαντές είναι ένα πεδίο Ισλαμικού φονταμεταλισμού και θα πρέπει να ελεγχθούν αυτά τα τζαμιά εκεί με ντρεσέντες. Αλλά η κυβέρνηση δεν ε, κάνει τίποτα για αυτούς τους εγκληματίες. Ε, και δεν κάνει τίποτα βεβαίω για να εκοσμικεύσει το κράτος και την κοινωνία. Εμείς λοιπόν συγγραφείς ε, δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε. Τα βιβλία μου απαγορεύονται, λογοκρίνονται και στον Παγκλαντές και στην Ινδία επειδή λέω την αλήθεια. Ε, αν ασκήσει κανείς κριτική τι χριστιανισμό, τον Ιουδαϊσμό, τον Ινδουισμό σε λένε διαφωτισμένο. Αν ασκείς κριτική στο Ισλάμ σε λένε Ισλαμοφοβικό. Και δεν θέλει κανείς να τον πούν ε, Ισλαμοφοβικό, οπότε το βουλώνει. Αλλά πώς πότε θα το βουλώνουμε. Οπότε αν θέλουμε να αλλάξουν οι μουσουλμανικές χώρες και οι κοινωνίες πρέπει να σκούμε κριτική στις ε, δογματικές πρακτικές του Ισλάμ. Οπότε κάτι που είναι αδύνατον στις μουσουλμανικές χώρες. Το Μπαγκλαντές ήταν κάποτε κοσμική χώρα, αλλά γίνεται Ισλαμική, φονταμεταλιστική. Το Πακιστάν ξέρετε πως είναι Ισλαμική φονταμεταλιστική χώρα. Οπότε εμείς όσοι πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα δικαιώματα των γυναικών, ε, το κοσμικό κράτος και τη δημοκρατία, υποφέρουμε. Δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε, αλλά σας ζητώ να κάνετε κάτι. Για να μπορέσουμε και να κάνουμε ε, τη δουλειά μας εκεί πέρα. Δεν θέμε να μας συλλαμβάνουν, να μας σκοτώνουν, δεν σκοτώσαμε εμείς κανέναν. Μιλάμε απλά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί μας σκοτώνουν γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Um, yes, I wait some uh, questions from... Πρόεδρος, μάλιστα. Υπάρχουν ερωτήσεις, σχόλια. Um, no sé si alguien ha levantado la mano, ¿no? Δεν βλέπω κανένα να σηκώνει το χέρι. Ο κύριος Αστρεβίσιος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε και μας ε, μιλήσατε για πράγματα τα οποία στην ουσία ε, μας δείχνουν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται. Αυτή η ατμόσφαιρα της ε, έλλειψης ανοχής είναι τόσο βαθιά ριζωμένη Ποια είναι η αντίδραση των ε, της, της κοινωνίας των πολιτών ε, των, όταν ας πούμε δολοφονούνται οι bloggers από ε, ακρο, ακραίους υπάρχει μια αντίδραση από την κοινωνία μια γενική αντίδραση παρατηρείται να αντιδράει η κοινωνία σε όλα αυτά Uh, Εγώ πιστεύω πως ο κόσμος φοβάται να στηρίξει τους ε, bloggers που είναι υπέρ της κοσμικότητας. Στο Μπαγκλαντές η λέξη άθεος είναι πολύ κακή λέξη. Κανείς δεν θέλει να υποστηρίξει λοιπόν έναν άθεο είναι ε, όλοι θρησκευόμενοι και οι άθεοι θα πρέπει να δολοφονούνται. Δεν υπάρχει καμία διαμαρτυρία κατά αυτών των δολοφονιών από πλευράς της κοινωνίας. Οπότε η κυβέρνηση, πιστεύω, γι' αυτό και η κυβέρνηση δεν προβαίνει σε ενέργειες κατά αυτών των δολοφόνων. Αλλά Από την άλλη δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμος δεν υποστηρίζει αυτούς τους blogger που δεν δολοφόνησαν ποτέ κανένα, δεν σκότωσαν ποτέ κανέναν, ούτε ε, διαπράξαν κανένα έγκλημα. Δεν δολοφονήθηκαν απλά και μόνο επειδή εξέφρασαν τη γνώμη τους που είναι διαφορετική από αυτή των φανατικών Φοβάμαι πως η Ισλαμοποίηση έρθει στα τέλη του 70 στον Παγκλατές Πάρα πολλοί κόσμος στράφηκε στη θρησκεία και στον εκτρεμισμό. Όχι, δεν γίνανε όλοι τρομοκράτες, αλλά κατά κάποιο τρόπο στηρίζουν την τρομοκρατία. Πολλοί κόσμος υποστηρίζει το ίσις και την Πόκο Χαράμα Και ε, άθεοι bloggers ε, ε, δολοφονούνται από τους Ισλαμιστές και οι απλοί μουσουλμάνοι στηρίζουν αυτές τις δολοφονίες. Είναι μια παράδεκτη κατάσταση, αλλά συμβαίνει λόγω αυτών των αλλαγών που έχουν γίνει στο Μπαγκλαντές. Δηλαδή ο φονταμενταλισμός έχει αντικαταστήσει το κοσμικό κράτος. Υπάρχει σύγκρουση όχι ανάμεσα στο χριστιανισμό και το Ισλάμ ή τον Ινδουισμό και το Ισλάμ. Η σύγκρουση είναι ανάμεσα στον φονταμεταλισμό και την, το κοσμικό κράτος ανθρωπισμός ε, έναντι βαρβαρότητος ε, ανάμεσα στο ανεκτικό και ε, κοσμικό κράτος και τη δικτατορία στην ουσία, αυτούς που εκτιμούν την ελευθερία και αυτούς που όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία... Ο κύριος Πανζέρη, με συγχωρείτε. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ δύσκολο να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. ενώπιον αυτού του αιτήματο που μας υποβάλλεται, τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει και δυσκολία από πλευράς μας να μπορέσουμε να ε, παρέμβουμε σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση από αυτή του Μπαγκλαντές, λαμβάνοντας υπόψη ότι και το Ευρωκοινοβούλιο επανειλημμένως έχει εκφράσει με διάφορα ψηφίσματά του ε, τη γνώμη του και έχει καλέσει την προσοχή της διεθνούς κοινή γνώμης ε, στη δύσκολη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαγκλαντές. Και ομολογώ ότι το θέμα της, κοσμικότητας και της ε, Ισλαμικής θρησκείας ε, είναι πολύ δύσκολο γιατί αυτό δεν προκύπτει από την ίδια τη θρησκεία όπως ε, προέκυψε από τη χριστιανική θρησκεία. Πολύ δύσκολο να έχουμε αυτή τη διάκριση των εξουσιών ανάμεσα στην πνευματική εξουσία και την χρονική εξουσία, την κοσμική εξουσία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι δυνατόν να κάνουμε στον Μπαγκλαντές, γιατί υπάρχει ε, οικονομική πίεση απέναντι στη κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, ε, επειδή ώστε μάλλον να υπάρξει πίεση οικονομική και ίσως θα μπορούσαμε να, να ενεργοποιήσουμε, δεν ξέρουμε τι, πώς, να ενεργοποιήσουμε μια συζήτηση στο πλαίσιο της ίδιας της αντιπροσωπείας της κοινοβουλευτικής για τις σχέσεις με την ε, Ινδία, ώστε να πιέσουμε και την Ινδία που έχει αντικειμενικά επιρροή στον Μπαγκλαντές και να μπορέσουμε έτσι να ε, ορίσουμε σαφέστερες ε, και να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες. Ε, αυτός θα ήταν ένας τρόπος για να μπορέσουμε λοιπόν να προχωρήσουμε μετά από τη σημερινή σας παρουσίαση να κάνουμε κάτι ώστε να κινηθούν τα πράγματα που αντικειμενικά η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Να ενεργήσουμε λοιπόν στο οικονομικό επίπεδο μέσω της Συμφωνίας Συνεργασίας καλώντας ε, να αναλάβει τις ευθύνες της κυβέρνησης κυβέρνηση του Μπαγκλαντές και από την άλλη πλευρά να δράσουμε ε, απέναντι στην Ινδία που είναι τόσο σημαντικός εταίρος του Μπαγκλαντές και που μπορεί να επηρεάσει και τις δράσεις της ε, κυβέρνησης του Μπαγκλαντές. Δώσω το λόγο στην κυρία Τόμασιτς και μετά στην κυρία Τεναστρίνη για να απαντήσει ώστε να διαβάσουμε και το γράμμα του κ. Σμάν που δεν μπόρεσε να έρθει μετά. Γεννήθηκα σε κομμουνιστική χώρα και γνωρίζω πως λειτουργεί ο κομμουνισμός ο κόσμος θεωρεί ότι αν παρακολουθείς ε, κάποιους άλλους τότε προστατεύεις ε, το ίδιο το κράτος οπότε καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους να ζουν στο Μπαγκλαντές. Έχω ένα ερώτημα. Ε, τι πιστεύετε ότι περιμένει ο λαός του Μπαγκλαντές από τη Δύση και τι μπορεί να κάνει η Δύση για να βελτιώσει την κατάσταση. Έχετε το λόγο. Αυτό ε, το οποίο ε, λένε οι κοσμικοί οι οποίοι απειλούνται από το Ισλάμ αφορά το ζήτημα της ασφάλειας. Θέλουν ασφάλεια στον Μπαγκλαντές, θέλουν να ζήσουν στον Μπαγκλαντές και να συνεχίσουν να έχουν τα δικαιώματά τους και ε, θέλουν η κυβέρνηση να μην, να μην ε, κινείται αρνητικά εναντίον τους αλλά εναντίον ε, των, των δολοφόνων, των φονταμελαζιστών, των ε, αυτών που τους απειλούν. Και τώρα εξαιτίας του φόβου ορισμένοι κοσμικοί blogger έχουν φύγει από τη χώρα όμως η κατάσταση δεν είναι τόσο εύκολη διότι αν φύγουν από τη χώρα τότε ποιος θα μείνει για να προσπαθήσει να αλλάξει την κοινωνία εκεί πέρα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φωτισμένοι και πρέπει να μείνουν στη χώρα και να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα ελεύθερης σκέψης στη χώρα. Θέλουν να έχουν ελευθερία έκφρασης. Είναι μια προσωρινή λύση το να βγουν από τη χώρα, όμως η μόνιμη λύση θα είναι να κατανοήσει η κυβέρνηση ότι οι φονταμενταλιστές δεν πρόκειται να κάνουν τη χώρα ένα καλύτερο μέρος. Ως δημοκρατική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές δεν θα πρέπει να παραβιέζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης. Αποτελεί αδύρυτη ανάγκη για τη δημοκρατία να έχει ελευθερία έκφρασης. Ορισμένες κυβερνήσεις ε, σε άλλες χώρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Μιλούν για δημοκρατία χωρίς όμως να πιστεύουν στην ελευθερία έκφρασης και με αποτέλεσμα να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν μπορέσετε λοιπόν να διδάξετε σε αυτούς τους πολιτικούς τη δημοκρατία τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάρτιν, θα μπορούσατε σας παρακαλώ να διαβάσετε το, την επιστολή του κυρίου Οσμάν ο οποίος ε, δεν μπορούσε να ταξιδεύσει από το Σουδάν εδώ πέρα και είναι η τρίτη φορά που του το απαγορεύουν αυτό. Είναι τιμή μου να διαβάσω την επιστολή του. Καταρχάς θα πω ότι τα αγγλικά δεν είναι μητρική του γλώσσα, οπότε θα το διαβάσω προσπαθώντας να διορθώσω κάποια ε, σημεία. Είναι, είναι ατυχές το ότι δεν μπορώ να παρευρεθώ στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχω ε, στο... Ε, στη συγκεκριμένη εκδήλωση διότι κατασχέθηκε το διαβατήριό μου όταν ταξίδευα προς, τις... προς τη Γενέβη. Παρ' όλα αυτά θα χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να επαναλάβω τα όσα είχα πει στο παρελθόν, στο χαρτούν αποτελεί ένδειξη της ε, πολιτικής της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης να αποστείλει τον ύπατο εκπρόσωπό της ε, δύο φορές στη Σουδία, στη, στο Σουδάν εκτιμώ την ανταπόκριση των αποστολών στις ανησυχίες και τα ερωτήματα. Θα επαναλάβω τα όσα είπα στην ομιλία μου. Πρώτον, το βασικό θέμα ανησυχίας είναι να προωθήσουμε πρωτοβουλίες για να σταματήσει ο πόλεμος μεταξύ της ε, κυβέρνησης του Σουδάν και των αντικαθεστωτικών που οδηγεί στον εκτοπισμό αμάχων ε, και αυτό οδηγεί σε αύξηση των προσφυγικών ροών μελλοντικά. Στο μέλλον η κυβέρνηση του Σουδάν θα πρέπει να επιτρέψει διεθνείς παράγοντες να έχουν πρόσβαση σε θύματα πολέμου χωρίς να έχουν κανένα περιορισμό και να έχουν δικαίωμα να παραμείνουν στα στρατόπεδα του IDP μέχρι να επιληθεί το ζήτημα. στα στρατόπεδα των εσωτερικά εκτοπισμένων. Θα πρέπει να υπάρξουν διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών και να έχει διαφορετική μορφή η διαπραγμάτευση αυτή από ό,τι στο παρελθόν. Δεύτερον, η κυβέρνηση του Σουδάν θεωρείται μια έξυπνη πλευρά που χρησιμοποιεί ζητήματα μετανάστευσης για να προωθήσει τα δικά τη συμφέροντα και σε αυτό το θέμα θεωρώ ότι η κυβέρνηση του Σουδάν έχει ως στόχο να προσκαλέσει και άλλους πρόσφυγες ε, στο Σουδάν μαζί και τρομοκράτες και τους χρησιμοποιεί ως ένα μέσο στη συνεργασία που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες απαιτώντας περαιτέρω συμβιβασμούς και άρση των κυρώσεων αλλά και χρηματική υποστήριξη. Εκατομμύρια θύματα γενοκτονιών θα απογοητευθούν εάν τους εγκαταλείψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τηρήσει τις αρχές της. Ιδιαίτερο όσον αφορά το ζήτημα της δικαιοσύνης. Τρίτον, οι άμεση παράγοντες οι οποίοι συμμετέχουν στο ζήτημα της Συρίας θα πρέπει να αλλάξουν ε, την πολιτική τους και να, πάρουν, να ακολουθήσουν βήματα για να κατοπολεμήσουν ε, την ε, μη επιβολή δικαιοσύνης και να επαναφέρουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και αυτό θα αποτελέσει διασφάλιση για την επιβολή δικαιοσύνης ε, για τα θύματα τα οποία επιζητούν ε, τη διεθνή δικαιοσύνη όταν ε, γίνεται παραβιάσεις, γίνονται παραβιάσεις και να γίνει δίωξη των υπευθύνων. Η δικαιοσύνη λοιπόν θα, θα βοηθήσει τις προσπάθειες για την ειρήνευση θα οδηγήσει σταθερότητα και περισσότερα θύματα θα θέλουν να παραμείνουν στα σπίτια τους από το να επιλέξουν την οδό της μετανάστευσης. Η αντικαθεστωτική είναι επίσης υπεύθυνη για τη συνέχιση του πολέμου, αρνούμενοι να συμμετέχουν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και παραβιάζουν τα δικαιώματα των μάχων και παραβιάζουν ταυτόχρονα τις συνθήκες ασφαλείας η διεθνής κοινότητα είναι υπεύθυνη για τη συνέχιση της ε, γενοκτονίας των Ταρφούν αλλά και τον εκτοπισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να αναθεωρήσει τις θέσεις της σχετικά με την υπευθυνότητά της πάνω στη γενοκτονία και να ακολουθήσει τις αξίες και τις αρχές της όσον αφορά τη συνεργασία με την κυβέρνηση του Σουδάν. Και τέλος, οι οργανώσεις ε, κοινωνίας των πολιτών θα μπορούν να παίξουν έναν θετικό ρόλο καλώντας όλες τις πλευρές να συμμετέχουν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με, ώστε να σταματήσει όχι μόνο ο πόλεμος αλλά και άλλα προβλήματα όπως είναι η παραβίαση της ε, ελευθερίας του λόγου και του συνεταιρίζεστε. Ελπίζω λοιπόν ε, να ε, επιτευχθεί αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάρτιν, λέει η Πρόεδρος. θα πρέπει να αποστείλουμε μια επιστολή και εμεί στον κύριο Όσμαν, ώστε να γνωρίζει ότι ακούσαμε τα λόγια του στην υποεπιτροπή μας, παρά το ότι δεν τον άφησαν να ταξιδέψει και ότι θα συνεχίσουμε να, προσπαθούμε να προσπαθούμε να το επιτραπεί το ταξίδι εδώ στη Βρυξέλλη, γιατί μου φαίνεται πως είναι άνθρωπος κλειδί στις σχέσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Σουδάν και όσον αφορά την εξέλιξη των ε, σχέσεων με αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ λοιπόν που μας διαβάσατε την επιστολή του κύριου Οσμαν. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Ναζρίν που ήταν εδώ μαζί μας. Να σας συγχαρώ όπως πάντα για την εργασία σας και για το θάρρος σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. y ahora eh, tienen... Eh, Και τώρα έχετε το εργαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα. Θα προεδρεύσει ο κύριος Τόκης. should start now. Yes. Please sit down, ladies and gentlemen. Παρακαλώ καθίστε, Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. στο σημερινό μας εργαστήριο που περιλαμβάνει μέλη της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε σήμερα τους ειδικού μας που θα μας βοηθήσουν για να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα για ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα όσον αφορά την λογοδοσία από πλευράς διεθνού κοινότητα για σοβαρέ παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε για την ε, λαοκρατική δημοκρατία της ε, Κορέας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον ε, Δ. Λί, πρέσβη για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Δημοκρατίας της Κορέας που ταξίδεψε από τη Σεούλ για να έρθει εδώ σήμερα αποφασίσαμε να οργανώσουμε αυτή τη συνεδρίαση για να αντιληφθούμε καλύτερα την κατάσταση και τις πολιτικές επιλογές που έχουν σχέση με την λογοδοσία για τις ε, σοβαρές και διαρκείς παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως ε, πραγματικά τα ευρήματα της Εξεταστικής Επιτροπής και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ ήταν, ε, είχαν ανεπανάληπτες διατυπώσεις. Μίλησαν για εκτεταμένα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν αλλού στο σύγχρονο κόσμο και ζήτησαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας να παραπέμψει το ζήτημα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Μάρτιο του 2016 ο ΙΕ αποφάσισε να συστήσει μια ομάδα ειδικών για να βοηθήσει περαιτέρω στο θέμα ακριβώ της λογοδοσίας. Ο κύριος Σαντάρσμαν, ο ειδικό ε, εισηγητής για τη Βόρεια Κορέα και μέλος της Εξεταστικής Αυτής Επιτροπής, δυστυχώς ε, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα είναι επίση πολύ ενεργό στο θέμα και είπε, πως η παρουσίαση της τελευταίας, είπε στην παρουσίαση της τελευταία του έκθεση πως η διεθνή κοινότητα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ηγεσία της Βορειας Κορέας και ειδικά ο κ. Κιμ θα πρέπει να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητα που διέπραξαν στη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως είναι το προσκήνιο όσον αφορά τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βόρεια Κορέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και υποστήριξε τη σύσταση μιας Επιτροπής Έρευνας θεωρεί πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πως πρέπει να ακολουθήσει μια πολιτική επικριτικής ε, εμπλοκής με την Βόρεια Κορέα. Δηλαδή αφενός έναν ε, πολιτικό διάλογο και κάποια προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας και από την άλλη στην διπλωματική πίεση και τις κυρώσεις. Οι πρόσφατες πυρηνικές δοκιμές και εκτοξεύσεις πυράβλων ε, είναι ανησυχητικές εξελίξεις για την ε, διεθνή κοινότητα. Και απειλούν να, να ε, αυξήσουν τις εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο παρά το ότι δεν έχει άμεση εμπλοκή στον τομέα της ασφάλειας η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει μια συνεχής ε, και αυξανόμενη ανάγκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν επικοδομητικό και ενεργό ρόλο. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρακολουθεί με ενδιαφέρον αυτό το θέμα, όπως ε, άλλωστε έδειξε και το ψήφισμα της 21ης Ιανουαρίου 2016 για την Βορεια Κορέα. Το ψήφισμα αυτό δηλώνει την ξεκάθαρη θέση μας για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει έναν επικοδομητικό ρόλο μέσω της ε, εμπλοκής αυτής που ανέφερα με την Βόρειο Κορεϊτική Κυβέρνηση. Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω πως ε, τον Οκτώβριο που μας πέρασε συστάθηκε η ομάδα Φίλιας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Δημοκρατίας Κορέας. Ε, ήμουν και εγώ μέλος υπό την προεδρία του κυρίου Ρούμπιχ. Ε, και είναι και ο, όπως είπαμε ο πρώτος πρόεδρος και έτσι έχουμε άμεσες επαφές με τον στρατηγικό αυτόν εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ασία για να προωθήσουμε ζητήματα αμοιβαίου συμφέροντος όπως το εμπόριο, η έρευνα και η ανάπτυξη, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ασφάλεια. Θα ήθελα λοιπόν να προσκαλέσω και άλλους συναδέλφους να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα. Με ιδιαίτερη χαρά. Καλωσορίζω τώρα την πρώτη ομιλήτρια, την κυρία Βερόνικα Μπίλκοβα, η οποία είναι ερευνητής ε, στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων της Πράγας, ειδική στο Διεθνές Δίκαιο και μέλος της Επιτροπής της Βενετίας, έχει γράψει για τις διεθνείς κυρώσεις ε, την επιβολή του διεθνούς ε, δικαίου. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Βόρεια Κορέα σε μια πρόσφατη μελέτη της με τίτλο «Ευθύνη προστασίας ε, πέρασμα στην Ευρασία και συγκεκριμένα θα μας πει πώς η διεθνή κοινότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στην διάθεσή της για να υπάρξει λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα τα θέσει αυτά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Σας παρακαλώ λοιπόν κυρία Μπίλκοβα. Έχετε τον λόγο. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μου δίνεται αυτή η ευκαιρία να σας απευθύνω το λόγο. Μου ζητήθηκε να επικεντρωθώ στους μηχανισμούς υπευθυνότητας όσον αφορά λογοδοσίας ε, σχετικά με την Βόρεια Κορέα και η ομιλία μου θα αποτελήσει μια εισαγωγή ε, για τις ομιλίες που θα ακολουθήσουν. Αρχικά θα σας δώσω ένα ε, υπόβαθρο ε, της κατάστασης και στη συνέχεια θα επικεντρωθώ στους μηχανισμούς λογοδοσίας καθώς επίσης θα δώσω και μερικές προτάσεις. Το ζήτημα της λογοδοσίας όσον αφορά την ε, Βόρεια Κορέα έχει λάβει κεντρική θέση ε, στην διεθνή σκηνή ιδιαιτέρως όταν ε, αφού η Επιτροπή Έρευνας, όπως αναφέρθηκε, εξέδωσε την έκθεσή της. Η έκθεση επιβεβαίωσε ότι υπάρχει μια συστηματική, ευρεία και κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς ε, άνευ προηγουμένου στην Βόρεια Κορέα για αρκετά χρόνια. Αυτές οι παραβιάσεις αφορούν ένα εύρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την ελεύθερη μετακίνηση, την ελευθερία ε, έκφρασης ε, και το δικαίωμα στη ζωή. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι αρκετές από αυτές τις παραβιάσεις αποτελούν ε, αδικήματα κατά της ανθρωπότητας. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ως αποτέλεσμα να απαιτείται η ευθύνη και η λογοδοσία από την πλευρά του κράτους ε, αλλά και των ε, ηγετών της χώρας. Η διεθνής κοινότητα λοιπόν μαζί και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τουλάχιστον την πολιτική ευθύνη να διασφαλίσει το ζήτημα της λογοδοσίας στη Βόρεια Κορέα και να βοηθήσει το λαό της χώρας ή στο πλαίσιο της, ε, της υπευθυνότητας για προστασία. Και θα χαρώ ιδιαιτέρως να ε, αναφερθώ καλύτερα σε αυτό. Δεν είναι ξεκάθαρο όμως και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα τι θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας διότι όπως θα δούμε όλοι οι μηχανισμοί λογοδοσίας αλλά και τα μέτρα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας έχουν τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα ή ακόμα και κινδύνους και έτσι λοιπόν θα φτάσω στο κεντρικό σημείο της ομιλίας μου. Όσον αφορά τα μέτρα λογοδοσίας, επέλεξα να τα κατηγοριοποιήσω σε τρία ε, μέρη με βάση το βασικό σκοπό που αποσκοπούν τα συγκεκριμένα μέτρα. Και είναι τα τρία ζητήματα να καταστήσουμε υπεύθυνου ε, όσους έχουν παραβιάσει ανθρώπινα δικαιώματα, στη συνέχεια να βοηθήσουμε τα θύματα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της Βόρειας Κορέας και τρίτον να βελτιώσουμε τη γενικότερη κατάσταση της χώρας. Όπως βλέπετε η λογοδοσία έχει κεντρικό ρόλο σε αυτή την παρουσίαση. Θα περάσουμε λοιπόν στο πρώτο ε, θέμα των μέτρων έχουμε επικεντρωθεί μέχρι στιγμής σε αυτή την κατηγορία και ορθώς διότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε δικαιοσύνη. Αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα θα πρέπει ε, να διωχθούν. Επιπρόσθετα, η εμπειρία δείχνει ότι ίσως να είναι δύσκολο να επιτύχουμε δικαιοσύνη σε μια χώρα η οποία μπορεί ε, να, η οποία ε, έχει ένα φαινόμενο ε, όπου απουσιάζει η δικαιοσύνη και υπάρχει ακόμα και κίνδυνος εμφύλιας διαταροχής όπως έχουμε δει στη Συρία, στην Ιουγκοσλαβία και σε άλλες περιοχές. Αυτό είναι δυνατό να διώξουμε τους υπεύθυνους ε, για κατάφορη παραβίαση δικαιωμάτων του ανθρώπου ε, στη Βόρεια Κορέα είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε σε άλλες χώρες. Όμως καμία από αυτές τις εναλλακτικέ δεν έχει λειτουργήσει. Η Βόρεια Κορέα για πασιφανείς λόγους δεν έχει τη βούληση ε, να κινηθεί νομικά εναντίον των ηγετών της και κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να αλλάξει το εγγύς μέλλον. Ταυτόχρονα όμως ε, κάτι τέτοιο σε άλλες χώρες ε, μπορεί να είναι δύσκολο διότι δεν μπορούμε να ε, συλλέξουμε αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν, από ό,τι ξέρω, δεν έχουν υπάρξει διώξεις σχετικά με τη Βόρεια Κορέα μέχρι στιγμής. Στην έκθεση του 2014 η Επιτροπή Έρευνας πρότεινε δύο άλλες εναλλακτικές Πρώτον, τη δημιουργία ενός ε, μιας ad hoc, ε, ενός ad hoc δικαστηρίου, όμοιο με αυτά τα οποία έχουν υπάρξει για την πρώην Ιουγκοσλαβία και την Ρουάντα, ή δεύτερον, ε, την αποστολή του ζητήματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα ξεκινήσω με το ad hoc δικαστήριο, είναι μια εναλλακτική που κατά τη γνώμη μου δεν συνίσταται διότι πρώτον ίσως να είναι δύσκολο να ε, δημιουργηθεί ένα τέτοιο δικαστήριο δεδομένου του ότι μερικά, ε, μερικές χώρες μεταξύ αυτών και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν βλέπουν θετικά τη δημιουργία νέων τέτοιων δικαστηρίων. Επιπρόσθετα ακόμα και αν δημιουργηθεί ένα τέτοιο δικαστήριο θα αντιμετωπίσει τις ίδιες δυσκολίες που βλέπουμε σήμερα με τα εθνικά δικαστήρια. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν για αρκετά χρόνια το δικαστήριο να μην έχει κανέναν τον οποίο θα δικάσει. Και αυτό ε, θα αποτελέσει μια αρνητική εικόνα όχι μόνο για τις δραστηριότητες του αλλά και ε, για το έβρος του. Οπότε δεν το συστήνω. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα ε, αντιμετωπίσει τα ίδια, ε, τα ίδια προβλήματα, διότι ίσως είναι δύσκολο να βρεθεί ομοφωνία στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, για το θέμα αυτό και ακόμα κι αν παραπεμφθεί η υπόθεση, τώρα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα δυσκολεύεται να βρει πρόσβαση σε θύματα, σε θύτες και ούτω καθεξής και ισχύει ότι η εμπειρία το επιβεβαιώνει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του μονάχα εάν η ενδιαφερόμενη χώρα δεν αντιτίθεται την δίωξη όπως συμβαίνει στην περίπτωση αυτή τη στιγμή του Σουδάνου όπου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν τα πηγαίνει καλά. Πιστεύω λοιπόν ότι η παραπομπή στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα πρέπει να υποστηριχθεί για δύο λόγους. Πρώτον, για συμβολικούς λόγους, πιστεύω ότι η παραπομπή θα αποστείλει ένα σημαντικό μήνυμα και θα δείξει ότι η διεθνής κοινότητα όντως ανησυχεί σχετικά με τα όσα ε, συμβαίνουν στη Βόρεια Κορέα. Το άλλο είναι πρακτικό θέμα. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα μπορέσει να αρχίσει να συλλέγει ε, αποδείξεις που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ήδη έχει ασχοληθεί με το ζήτημα της Βόρειας Κορέας, όχι με την κατάσταση ε, την ίδια, αλλά με την Βόρεια Κορέα το 2014 ένα ζήτημα που αφορούσε ένα συνοριακό ατύχημα μεταξύ της Βορείου και της Νοτιού Κορέας και τότε αποφάσισε λοιπόν ότι τίποτα δεν ε, αποδείχνει πως έχει δικαιοδοσία σε αυτό το θέμα. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν είναι προκατηλημένο απέναντι στη Βόρεια Κορέα και αυτό είναι σημαντικό. Με βάση αυτές τις ε, εναλλακτικέ προτείνω την παραπομπή, όμως δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από αυτή την πρώτη κατηγορία μέτρων. Υπάρχουν κάποια τα οποία πρέπει να γίνουν την σωστή στιγμή, όμως αυτή η στιγμή μάλλον δεν έχει έρθει ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Τώρα περνώντας στην επόμενη κατηγορία των μέτρων λογοδοσίας, εδώ καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι την λογοδοσία με τη γενικότερη έννοια. Αυτή περιλαμβάνει μέτρα που θα πρέπει να παρέχουν άμεση βοήθεια στα θύματα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της χώρας. Σε αυτή την παρουσίαση σας δίνω τέσσερα παραδείγματα μια τέτοιας εναλλακτική μέτρων ε, και μηχανισμών, όμως σίγουρα υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Δύο σημαίνουν την παροχή υλική βοήθειας αλλά και την ε, παροχή πληροφόρησης που θα πρέπει να γίνεται στο εσωτερικό της Βόρειας Κορέας παρέχοντας άμεση βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται και ταυτόχρονα θα πρέπει να δίνονται εναλλακτικέ πληροφορίε για την κατάσταση στη χώρα. Τα μέτρα αυτά αφού εφαρμοστούν θα πρέπει να εφαρμοστούν πολύ προσεκτικά και η επιρροή τους αλλά και τα ρίσκα τα οποία συνδέονται είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα άλλα δύο μέτρα αφορούν την συνεργασία και είναι μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν έξω από τη Βόρεια Κορέα, ιδιαίτερα στις χώρες της περιοχής εκεί. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε ε, την ε, τακτική του non-refoulement για την Βόρεια Κορέα. διότι σε περίπτωση που επιστραφούν στην χώρα οι πολίτες αυτοί μπορεί να αντιμετωπίσουν κυρώσεις. Αποζημιώσεις είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο πολλοί το αντιλαμβάνονται ως χρηματικές αποζημιώσεις. Η δική μου κατανόηση είναι γενικότερη και περιλαμβάνει και ψυχολογική βοήθεια που θα παρέχεται στα θύματα, αλλά και προγράμματα ε, που θα τους βοηθήσουν να επανενταχθούν και αυτό ε, μπορεί να γίνει στο εξωτερικό της χώρας και υπάρχει βέβαια υποχρέωση των χωρών να παρέχουν τέτοια βοήθεια ακόμα και σε θύματα ε, παραβιάσεων που έχουν προκληθεί από άλλους. Αυτά τα δύο μέτρα λοιπόν ε, χρειάζονται διεθνή ε, συνεργασία διότι οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν ε, στην, που παραμένουν στη χώρα χρειάζονται αυτά τα μέτρα. Η εφαρμογή όμως μπορεί να προωθηθεί από το εξωτερικό και ιδιαίτερα στα μέτρα αποζημιώσεων μπορούν να συσχετηθούν με κάποια χρηματική βοήθεια από το εξωτερικό, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράδειγμα. Φυσικά τα μέτρα αυτά δεν είναι καινούργια, έχουν εφαρμοστεί, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που προτείνω. Όμως το καινούριο είναι ότι δεν, έχουν, δεν τα έχουμε αντιληφθεί ως μέτρα λογοδοσίας και θεωρώ ότι θα πρέπει να αντιληφθούμε έτσι. Και το ίδιο ισχύει και για την τελευταία κατηγορία μέτρων, τα οποία είναι πιο γενικά και έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα. Υπάρχουν τρία, ε, τρία είδη μέτρων διπλωματικά εργαλεία, πολιτικά εργαλεία, στοχευμένες κυρώσεις και τέλος θεωρητικά η χρήση ε, του στρατού. Λέω θεωρητικά διότι δεν πιστεύω ότι μια στρατιωτική επέμβαση στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το επιτύχουμε. Η κίνδυνη ε, είναι πολύ υψηλή τόσο για τους κατοίκους όσο και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειε για αυτό, νομίζω ότι είναι πασιφανέ. Οπότε έχουμε τα πολιτικά εργαλεία και τι ε, κυρώσει. Τα πολιτικά εργαλεία περιλαμβάνουν διάλογο με την ίδια τη Βόρεια Κορέα, με άλλε χώρε, καθώ επίση και την ενεργητική χρήση ορισμένων μηχανισμών του ΟΗΕ όπως είναι για παράδειγμα ε, εκθέσεις, ε, παρατηρητές ε, με θεματική εντολή ή με βάση τη χώρα καθώς επίσης και μια ομάδα ειδικών που προαναφέρθηκε τα συγκεκριμένα πολιτικά εργαλεία μπορεί να μην θεωρούνται ιδιαίτερα αυστηρά και ίσως είναι δύσκολο να διασφαλίσουμε ε, διάλογο για σημαντικά ζητήματα όπως είναι η πολιτική κρατούμενη ή η ελευθερία έκφρασης για τον απλούστατο λόγο ότι η Βόρεια Κορέα αρνείται ότι υπάρχουν τέτοιοι κρατούμενοι όμως ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τα συγκεκριμένα μέτρα και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερως κατά τα τελευταία χρόνια η Βόρεια Κορέα έχει δείξει βούληση να ξεκινήσει διάλογο με τους μηχανισμούς του ΟΗΕ το 2008 αλλά και το 2014 έλαβε ενεργό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο και αυτό δείχνει ότι ίσως να έχει τη βούληση να αποδεχθεί τις περισσότερες προτάσεις. Αυτό για την πρώτη κατηγορία. Τώρα όσον αφορά τις στοχευμένες κυρώσεις, η Βόρεια Κορέα υπόκειται κυρώσεις εδώ και πάρα πολύ ε, καιρό, όπως ε, σημείωσε η Επιτροπή Ερευνών όμως, οι συγκεκριμένες κυρώσεις δεν είναι στοχευμένες και αυτό πρέπει να αλλάξει, διότι ε, δεν θέλουμε να βάλουμε τους απλούς πολίτες αλλά την ηγεσία. Θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα λοιπόν το ζήτημα των στοχευμένων κυρώσεων και τέλος κάποιες γενικές προτάσεις με τις οποίες θα ήθελα να ολοκληρώσω. Ο τελικός στόχος λοιπόν όλων αυτών των μέτρων λογοδοσίας είναι και θα πρέπει να είναι να βοηθήσουμε τον πληθυσμό της Βόρειας Κορέας Θα πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε όλο πολύ προσεπτικά. Τα μέτρα δεν πρέπει να κάνουν μεγαλύτερο κακό ε, και αυτό ισχύει στην περίπτωση της στρατιωτικής επέμβασης. Δεύτερον, όλα αυτά τα μέτρα λογοδοσίας θα πρέπει να στοχεύουν στους τρεις στόχους. Ε, λογοδοσία των υποθήνων, να βοηθήσουμε τα θύματα και να βελτιώσουμε τη γενικότερη κατάσταση. Αυτή οι στόχοι είναι αλληλοσυνδεδεμένοι, είναι εξίσου σημαντικοί, όμω δεν μπορούν να επιτευχθούν κατά πάσα πιθανότητα ταυτόχρονα και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η κατηγορία 2 και 3 θα πρέπει να έχει προτεραιότητα για την ώρα. Τρίτον, δεν υπάρχει μία ε, λύση ως εκθαύματος, ε, ως εκθαύματος. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε σε έναν συνδυασμό διαφορετικών μέτρων όπως ανέφερα Χρειαζόμαστε επίσης, και αυτό ίσως να ακουστεί εξοργιστικό, χρειαζόμαστε υπομονή, διότι τα μέτρα αυτά δεν πρόκειται να φέρουν αλλαγή εν μία νυχτή. Και τέταρτον, τέλος, Ευχαριστώ. Ναι, ζητώ Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη ε, που σας διέκοψα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με τον επόμενό μας ομιλητή, που είναι ο, ο δόκτωρ Πατσέκο Πάρτο. φυγητής Διεθνών Σχέσεων στο King's College του Λονδίνου. Βασικός τομέας έρευνας και διδασκαλίας του είναι οι σχέσεις Ένωσης Ανατολικής Ασίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ε, Κορεατική Χερσόνησο. Ο Δ. Πατσέκο Πάρτο έχει κάνει διάφορες εισηχήσεις για αυτές τις πολιτικές σε ακροατήρια ε, ε, και επίσης συμβάλλει τακτικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ανατολικής Ασίας. Διεξάγει έρευνα για τη Βόρεια Κορέα και τους νέους φόβους ε, για την κορεατική ε, ε, Χερσόνησο καθώς και σε σχέση με το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας καθώς και σε σχέση με την μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Επίσης, εξετάζει την ένταξη της Βόρειας Κορέας στις παγκόσμιες προσπάθειες για τη βελτίωση των, της διαβίωσης των Κορεατών. Ο Δ. Πατσέκο θα μας μιλήσει για το δύσκολο θέμα της ε, ε, εμπλοκής με τον DPRK το, το, το πώς θα μπορέσει η διεθνής κοινότητα να επηρεάσει, το πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε την ανθρωπιστική βοήθεια, τις οικονομικές εξελίξεις, κυρώσεις, ποινές και άλλες διεθνείς προσπάθειες όσον αφορά την μη εξάπλωση των πυρηνικών. Κύριε Πατσίκο Πάρντο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόκληση, η πρόσκληση να μιλήσουμε για τα θέματα για το, ε, σε επαφέ με τη Βόρεια Κορέα που είναι κλειδί εάν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Βόρεια Κορέα και να ε, συμβάλλουμε στην οικονομική μεταρρύθμιση και ίσως ποιος ξέρει και την πολιτική μεταρρύθμιση της χώρας. Εγώ θα εστιάσω σε τέσσερα διαφορετικά θέματα, πολύ σύντομα. Ποια είναι τα βασικά ε, επιχειρήματα που παρουσιάζει η Βόρεια Κορέα και πώς μπορούμε να αναχαιτήσουμε. Μετά θα εστιάσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική δέσμευση, τα οικονομικ... τους οικονομικούς μηχανισμούς που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορούσε ίσως να τους χρησιμοποιήσει με διαφορετικό τρόπο, πολιτική εμπλοκή και μετά θα προβώ σε συστάσεις. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μοναδική στις σχέσεις ε, με την Βόρεια Κορέα. Όλο είναι και περισσότερο θεωρείται αξιόπιστος εταίρος ως ένας ε, εταίρος που θέλει να εφαρμόσει οικονομική και διπλωματική εξουσία χωρίς να έχει όμως δυτική παρουσία που είναι βασική διαφορά από άλλες χώρες που ενδιαφέρονται για τα θέματα της Βόρειας Κορέας αλλά επίσης θεωρείται και ως ένας ειλικρινής διαμεσολαβητής γιατί δεν έχει στρατιωτική παρουσία η εξωτερική της πολιτική δεν περιλαμβάνει στρατηγικά στοιχεία που περιλαμβάνουν οι στρατηγικές των ΗΠΑ ή της ε, Ρωσίας. Μπορεί λοιπόν να παίξει και ε, σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ποια είναι τα επιχειρήματα της Βόρειας Κορέας ε, Καταρχά μιλά για την πυρηνική αποτροπή, γιατί λέει ότι είμαστε ακόμα σε εμπόλεμη κατάσταση, ότι αυτή τη στιγμή ισχύει η ανακοχή που υπογράφηκε μετά τον πόλεμο τη Κορέα ε, το 1953, αλλά δεν υπάρχει ε, συνθήκη ειρήνη. οπότε πρέπει να μπορούμε να αμυνθούμε, δεν γίνεται κανένα διάλογο με τι χώρε Και τελευταία στοιχεία, και το άκουσα αυτό από πρέσβεις της Βόρειας Κορέας και επισήμους, λένε τα η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετίζεται με το γεγονό ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και πρέπει να προστατεύσουμε τη χώρα μα από του εσωτερικού εχθρού. Αυτό λέει η Βορειοκορεάτε. Χρειαζόμαστε σταθερότητα. Οι οικονομικέ κυρώσει είναι ω ένα εργαλείο, ω ένα πόλεμο κατά τη Βόρεια Κορέα και οι οικονομικέ μεταρρυθμίσει που έχουν ξεκινήσει από το 2002 στη χώρα είναι, ε, στόχο έχουν να βελτιώσουν αλλά όχι να αλλάξουν το ισχύον κοινωνικό σύστημα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλήσουμε με τη Βόρεια Κορέα με τους δικούς της όρους. Αυτό όλα βέβαια συνάδουν στο γεγονός ότι αυτή η χώρα αισθάνεται απομονωμένη, παρεξηγημένη και επίσης ε, αισθάνεται και προσβεβλημένη γιατί η Νότια Κορέα είναι πολύ πιο επιτυχημένη η χώρα ε, και έχει χάσει έτσι η Βόρεια Κορέα τον ιδεολογικό πόλεμο, τον ιδεολογικό αγώνα στην κορετική Χερσόνησο. Τώρα εστιάζουμε στην οικονομική τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν αλλάξει τη συμπεριφορά της η Βόρεια Κορέα και τι μπορεί να κάνει αν Όντω η χώρα αυτή θελήσει να συνεργαστεί περισσότερο. Και το λέω αυτό γιατί αν δούμε τη συνεργασία τη βόρεια κορέα με τον υπόλοιπο κόσμο, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου είχαμε διμερεί ε, διαπραγματεύσει με την Νότια Κορέα, είχαμε τετραμερείς συνομιλίε, εξαμερείς συνομιλίε, είχαμε ε, μια ε, οργάνωση για την ανάπτυξη τη χερσονήσου τη Κορέα, δηλαδή κάποια φάση θα πρέπει να υπάρξει η επανάληψη βιώσιμων σχέσεων με την Βόρεια Κορέα και αυτό πρέπει να το Εάν δεν αλλάξει η συμπεριφορά τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να έχει μια βοήθεια, ένα πρόγραμμα βοήθειας με βασικό γνώμονα την ε, απόπειρα για βελτίωση τουλάχιστον μάλλον για την αποφυγή λοιμού, όπως είχαμε το 1990, αν όχι τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Βορειοκορεατών. Θα μπορούσαμε όμως να έχουμε τέτοιου στόχου γιατί η Βόρεια Κορέα λέει για παράδειγμα ότι θέλει να βελτιώσει την ε, βιομηχανία τουρισμού της. Ε, ότι έχουμε εκείνο το, το, το ηφαίστειο, πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πιθανή έκρηξη του ηφαιστείου στη Βόρεια Κορέα. Δηλαδή υπάρχουν ανοίγματα ε, που πρέπει να τα δούμε ε, αυτά, ως, όχι άμεσα βέβαια ως ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πάντως ως στοιχεία που θα βελτιώσουν τη διαβίωση των Βορειοκορεατών που μπορεί να μην ε, μπαινούν, να μην είναι μέση τάξη. Ας πούμε οι επιστήμονες ή αυτοί που εργάζονται στο τουριστικό τομέα, αλλά αυτή τη στιγμή αυτά όλα παραμελούνται λόγω μέσω μάλλον τη ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε καλύτερα να συντονιστεί με άλλου εταίρους. Ακριβώ επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εδώ και πολύ καιρό συνεργαστεί χωρί διακοπή. Η για παράδειγμα κάποιε φορέ αλλάζουν πολιτική, σταματούν, κάποιε φορέ ε, μπλέκονται, κάποιες... με την Ιαπωνία το ίδιο συμβαίνει, η Νότια Κορέα είναι άλλη υπόθεση. Ε, πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει συντονιστικό ρόλο ακριβώς επειδή θέλει να συνεχίσει με αυτήν την δέσμευση που έχει απέναντι, στη, αναλάβει, απέναντι σε αυτή τη χώρα και αυτό και με τις προσπάθειες για την μη εξάπλωση των ε, ε πυρηνικών. Θα μπορούσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εκφράσει τις ανησυχίες αυτές όλες προς την χώρα. Τέλος, πιστεύω μακροπρόθεσμα ότι σε 5-10 χρόνια θα πρέπει να εξετάσουμε τη δυνατότητα ανάληψης ε, δράσης βήμα προς βήμα, όπως ε, αυτοί που συμφώνησαν οι εξαμερείς συνομιλίες το Σεπτέμβριο του 2005. Ε, εκεί είχε συμφωνηθεί μια ξεκάθαρη προδιαδικασία σε φάσεις όπου κάθε δράση θα έπρεπε να παίρνει και απάντηση από τη Βόρεια ε, Κορέα. Ίσως λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να το εξετάσει στο μέλλον, αν δεν υπάρξει αλλαγή συμπεριφορά. Τώρα, αν υπάρξει αλλαγή συμπεριφορά και χθε, για παράδειγμα, ε, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΕΠΑ ε, είπε ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με το Βόρεια Κορέα όπως με την Κούβα ή το Ιράν. Μπορεί να συμβεί αυτό και μάλιστα το βρίσκω πολύ πιθανό. Projects δηλαδή που είναι πολύ σημαντικά για την οικονομική ανάπτυξη της Βόρειας Κορέας θα μπορούσαν να συνδεθούν σαφώς με την σταδιακή μείωση ε, της εξάπλωσης των μέσων μαζικής καταστροφής, των πυρηνικών όπλων δηλαδή, και αυτό μέσα σε μια πορεία βήμα-βήμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ρόλο κλειδί, μπορεί να παρέχει την δυνατότητα κατάρτισης, εκπαίδευσης ε, και δημιουργίας δυνατοτήτων έτσι ώστε λόγω μάλλον των ε, πολιτών, της πολιτούς της δέσμευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει στο παρελθόν, αλλά διακόπησαν τα προγράμματα αυτά. Και η Αυστρία, ας πούμε, το έχει κάνει αυτό. Στη Σιγκαπούρη υπάρχει οργάνωση που προσπαθεί να το κάνει αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως πιστεύω πως έχει περισσότερες δυνατότητες να το καταφέρει. Μέσω πρόθεσμα επίσης εστιάζουμε στα ανθρώπινα, ανθρώπινα δικαιώματα. Α, αν δούμε το Σύνταγμα της Βόρειας Κορέας, υποτίθεται ότι είναι ο παράδεισος του εργαζομένου, του εργάτη. Ωραία λοιπόν. Γιατί να μην βελτιωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν θέλησαν να το συζητήσουν. Υπάρχουν χιλιάδες ε, Βόρειο ε, στο εξωτερικό που δουλεύουν σε πολύ άσχημες συνθήκες. Αν μπορούμε να το, να το επηρεάσουμε αυτό, μπορούμε να ξεκινήσουμε με ευρωπαϊκά προγράμματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Να ενημερώσουμε γι' αυτά και σιγά σιγά να προχωρήσουμε και σε άλλα θέματα. Να μιλήσουμε για ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα και τις φρικαλαιότητες που ε, διαπράττονται κατά του πληθυσμού της Βόρειας Κορέας. Βέβαια, τις τελευταία 10 χρόνια η Βόρεια Κορέα άλλαξε βιολή. Μιλούσε, πριν από 10 χρόνια δεν μιλούσε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τώρα τουλάχιστον μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα, οπότε ας μιλήσουμε μαζί τους για αυτά που θέλουν να συζητήσουν. Όπω και με οποιαδήποτε άλλη χώρα, υπάρχουν κομμάτια που θέλουν να ανοίξουν. Συνέβη τα 70, τη δεκαετία του 70 στην Κίνα, στο Βιετνάμ τη δεκαετία του 90, συμβαίνει σήμερα στην Μιανμάρ. Ε, οπότε βλέπουμε διάφορες συνιστώσεις ε, ε, μέσα σε μια, μάλλον φατρίες, μέσα σε μια κυβέρνηση που έτσι Αυτές οι φατρίες εξαρτώνται όλο και λιγότερο από την κεντρική κυβέρνηση λόγω των πολύ κακών συνθήκων και μπορεί να είναι πιο πρόθυμες να ανοίξουν προς τα έξω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν ε, συμμετέχει σε πολιτικό διάλογο με την Βόρεια Κορέα. Υπήρχε και ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει τώρα διακόπη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πάντως αυτό που πιστεύουμε ότι είναι μοναδικό είναι πως αυτός ο διάλογος συνεχίζεται εδώ και 15 χρόνια και παραπάνω στα τέλη της δεκαετίας του 90 χωρίς διακοπή. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν με αυτό το πολιτικό διάλογο. Πρώτον, να καταστήσουμε σαφέ στη Βόρεια Κορέα ότι αυτό ο διάλογος θα διατηρηθεί, αλλά ότι θα, θα είναι κομμάτι του και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να επιμένουμε σε αυτό. Η μη εξάπλωση επίση είναι ανησυχία τη Διεθνή Επιτροπή και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. τα ανθρώπινα δικαιώματα, λοιπόν, αν, είδαμε α πούμε τη δεκαετία του 80 και του 90 στην Κίνα Είχαμε πολύ ισχυρό διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως να θελήσουν και εκείνοι να το ε, συζητήσουν. Μπορούμε επίσης να δούμε ε, ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής για, για τις χώρες που δεν θέλουν να συνομιλήσουν απευθείας με τη χώρα αυτή. Και τέλος, και αυτό σχετίζεται και με αυτά που είπα προηγουμένως για την οικονομική εμπλοκή, η ιδέα της εξοικείωση με τους κυβερνητικού εκπροσώπους. Έχουμε ερευνητικά προγράμματα, έχουμε, ε, αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με το πολιτικό διάλογο και να βελτιωθεί μέσω περισσότερης δέσμευσης ε, από πλευρά τη Ένωση, ώστε να αγγίξουμε κόσμο που δεν θα αγγίζαμε μέσω του πολιτικού διαλόγου. α πούμε, αναφέρα τον τομέα του τουρισμού, όπου υπάρχει ένα θεσμό ε, στην Ολλανδία που τώρα βοηθά την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας να αναπτύξει το τουριστικό τομέα μέσω του, ας πούμε, της κατάρτισης τουριστικών ξεναγών. Εάν δεν αλλάξει. Μάλλον, αλλάξει μάλλον η συμπεριφορά της Βόρειας Κορέας και θελήσει να συνομιλήσει με το διάφορο, και με άλλους εταίρους εκτός από την Ένωση. Οι διάφοροι διάλογοι είναι καλό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μιλάει για κάτι και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συνομιλεί και να αναγνωρίζει τις ανησυχίες της χώρας. Και το αναφέρω αυτό ε, γιατί ε, είπε η συνάδελφος ότι η Βόρεια Κορέα αισθάνεται απομονωμένη. Αλλά όταν ας πούμε μιλάμε με πανεπιστημιακούς της χώρας ή μπορούμε να είναι διαφορετικά τα πράγματα ή μπορεί να μιλήσουμε με ε, μέρη της κυβέρνησης ε, ή διοικητικούς υπαλλήλους, να δούμε δηλαδή πώς θα εκπαιδεύσουμε τον πληθυσμό της Βόρειας Κορέας ώστε να, οδηγήσει σε μια, να οδηγηθεί μάλλον σε μια ευημερή οικονομία, κάτι που έχει αποτύχει μέχρι στιγμής. Ε, επίσης θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, όπως είπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτόν τον τρόπο, αλλά να διευκολύνουμε και τον ε, ατομικό προσωπικό διάλογο με άλλες χώρες οι προσωπικές επαφές δημιουργούνται μόνες τους, αλλά με τη Βόρεια Κορέα υπάρχει τόσο έντονος έλεγχος στην κοινωνία που η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει τα δικά της και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιμείνει περισσότερο για την ανάγκη να ξεπεράσουμε τους ε, κυβερνητικούς εκπροσώπους και να συνδεθούμε με άλλους ανθρώπους, πράγματα που μπορούν να γίνουν μέσω της παιδείας και των ερευνητικών προγραμμάτων ε, όπως αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Τέλος, οικοδόμηση εμπιστοσύνη και εξοικείωση με τους κυβερνητικούς υπαλλήλους ε, της Βόρειας Κόρεας, ε, ανώτερο επίπεδο αλλά και σε κατώτερο επίπεδο, δηλαδή τον κόσμο που θα παίξει ρόλο στην Βόρεια Κορέα. Αυτό λειτουργήσε πολύ καλά στην ε, Κίνα και στο Βιετνάμ. Αυτή είναι η εντύπωσή μου. Με την Μιανμάρ τώρα ξεκινάνε όλα αυτά και θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο και με τη Βόρεια Κορέα. Σύντομα, οι βασικές συστάσεις για την Ένωση και για το Ευρωκοινοβούλιο, ε, καταρχάς για την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουμε με τον τακτικό πολιτικό διάλογο, να μην το παραμελήσουμε, ακόμα και αν άλλε χώρες δεν είναι πρόθυμες να συνεχίσουν, ε, να βελτιώνεται η βοήθεια και η αρρωγή στη κοινωνία των πολιτών και θεσμοθέτηση των μηχανισμών αυτών, καθώς και συντονισμός με τους διεθνείς εταίρους, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην διεθνή κοινότητα και τη Βόρεια Κορέα. Τέλος, οι σχέσεις για το... Μάλλον, οι το ίδιο το Κοινοβούλιο, οι συστάσει προς το ίδιο το Κοινοβούλιο. Υπάρχει ομάδα εργασία στο Κοινοβούλιο για, για τη Βόρεια Κορέα. Από άλλε δεν έχουν καν κάνει κάτι τέτοιο. Τη δεκαετία του 70 η συνέλευση, η ανώτατη λαϊκή συνέλευση χρησιμοποιήθηκε από τη Βόρεια Κορέα για να προσεγγίσει το κογκρέσο, ε, το Αμερικανικό κογκρέσο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε εδώ. Ε, να μην συζητήσουμε στα δικαιω... για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο κυβέρνηση. αλλά να συζητήσουμε για άλλα πράγματα όπως ε, η μη εξάπλωση και τέλος να υπάρξει συντονιστό με τους διεθνείς εταίρους, γιατί κατά τη γνώμη μου η, κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ισχυρέ ομάδε που μπορούν να ε, και έχουν, έχουν μάλλον εργαστεί στη Βόρεια Κορέα για 5, 10, 15, ακόμα και 20 χρόνια και μπορούν να βοηθήσουν ώστε να έχουμε μια καλύτερη προσέγγιση προς την ε, Βόρεια Κορέα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Pacheco Pardo. The following speaker will be Σας ευχαριστώ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Σίλβια Κατερίνη, σύμβουλος ε, του έργου λογοδοσίας της ε, Βορειάς Κορέας. Μία πρωτοβουλία που έχουν ξεκινήσει διάφοροι ενδιαφερόμενοι για να στηρίξουν τις προσπάθειες του ΟΗΕ για να υπάρξει λογοδοσία για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα μας μιλήσει για τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και την συνεισφορά τους ε, μαζί με τις διαδικασίες του ΟΗΕ μεταξύ των οποίων και η καταγραφή και η τεκμηρίωση των παραβιάσεων ανθρωπινών δικαιωμάτων, ε, η δουλειά που κάνουν με θύματα και ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν από την ε, Βόρεια Κυρία Σίλβια Κατερίνη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Σίλβια Κατερίνη και εκπροσωπώ το North Korean Accountability Project. Όπως ήδη υπόθηκε, πρόκειται για κάτι το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα μετά από προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών που ασχολείται με την Βόρεια Κορία. μετά από τις προσπάθειες όσων ξεκίνησαν την Εξεταστική Επιτροπή το 2013 και μετά από τα ευρήματα αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν κάποια βήματα για να λογοδοτήσουν οι ηγέτες ε, της ε, Βορείου Κορέας για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Υπάρχουν κάποια έγγραφα για το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε στην αίθουσα. Να κάνω όμως μια σύντομη εισαγωγή. Ο κύριος στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το διεθνές ε, πλαίσιο, να δούμε το τι μπορεί να γίνει για να λογοδοτήσουν οι ηγέτες και δεύτερον θα ζητήσουμε να γίνουν συγκεκριμένα βήματα και να κοιτάξουμε εντός ε, του πλαισίου του ΙΕ αλλά και παραπέρα για να δούμε το τι μπορεί να γίνει για να λογοδοτήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό θα γίνει μέσω τριών ε, αλληλένδετων ε, δράσεων. Πρώτα απ' όλα βεβαίως έρευνα. Να δούμε ποιες είναι οι επιλογές ε, για λογοδοσία στη Βόρεια Κορέα. Δεύτερον, θα γίνουν κάποιες διαβουλεύσεις και στήριξη των επιζώντων και των θυμάτων της Βόρειας Κορέας για να μπορέσουν έτσι να εκφράσουν τις απόψεις τους για το ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για την απόδοση δικαιοσύνης για τα δικαιώματα κατά της ανθρωπότητας ε, που ε, διεπράχθησαν στη Βόρεια Κορέα και βεβαίως ε, θα προσφέρουμε στήριξη για το πώς θα μπορέσουν να εφαρμοστούν οι συστάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής και βεβαίως θα είμαστε σε επαφή με την ομάδα ανεξαρτήτων ειδικών του ΟΗΕ που συστάθηκε τον Μάρτιο και θα έχει μια εντολή 6 μηνών από το Σεπτέμβριο του 2006 και μετά. Για να αντιληφθούμε λοιπόν πώς ξεκίνησε η δικιά μας η δουλειά θα πρέπει να σας δώσω μια γενική εικόνα του τι κάνουν οι ΜΚΟ και τι κάνει η κοινωνία των πολιτών ε, όταν μιλάμε για λογοδοσία. Στο ένα άκρο έχουμε ΜΚΟ όπως οι απαχθέντες ε, του πολέμου της Κορέας που ζητάνε από τον ε, Διεθνή Ερυθρό Σταυρό να κάνει έρευνες για τις απαγωγές Νότιο Κορεατών και επειδή έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης εμείς λέμε πως οι εξαφανίσεις αυτές είναι εγκλήματα και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Επίσης ξεκινήσαμε μόλις να μιλάμε για λογοδοσία. Αυτό ξεκίνησε αμέσως μετά την έκθεση της ε, Επιτροπής αυτής η οποία για πρώτη φορά όπως είπαμε μετά τις έρευνές της μίλησε για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ακριβώς λόγω αυτής της γκρίζα ζώνης μπορεί και ε, δραστηριοποιείται η οργάνωσή μας. Θεωρούμε όμως ότι στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας βλέπουμε ότι οι προσπάθειες ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, είναι σπάνιες και δεν έχουν σχεδόν κανένα νόημα, οπότε θα έπρεπε κάτι να γίνει. Αν οι αρχές της ε, Βόρειας Κορέας παραδεχτούν προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τότε θα άξιζε να υπάρξει κάποια εμπλοκή, αλλά πάντα βεβαίως χωρίς ανταλλάγματα για αυτή την λογοδοσία. Οπότε εμείς θεωρούμε πως αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι αλληλοαποκλείωμενα. Δηλαδή πρέπει να δούμε και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και την λογοδοσία. Το ερώτημα λοιπόν δεν θα έπρεπε να είναι το εάν θα υπάρξει λογοδοσία, αλλά πώς θα γίνει αυτό και πότε. Το διεθνές δίκαιο απαιτεί οι υπεύθυνοι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας ε, να λογοδοτούν και η διεθνής ε, κοινότητα έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει για να αντιληφθούν οι χώρες ε, πως υπάρχει μια υποχρέωση να αντιδράσουν όταν διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι στην Ιρεμβέργη, στην Καμπότζη, μετά την γενοκτονία της Ρουάντας και το ερώτημα είναι πως θα υπάρξει κάποια δίωξη αυτών των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Βεβαίω η περίπτωση της Βόρειας Κορέας είναι κάτι το άνευ προηγουμένου ε, και έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Ε, όμως ε, θεωρούμε πως η άνευ προηγουμένου βαρβαρότητα και το ότι τα εγκλήματα αυτά διαρκούν ε, γενιές ήδη ε, σημαίνει ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απόδοσης δικαιοσύνης. Εμείς θεωρούμε λοιπόν πως τώρα θα πρέπει να εστιάσουμε στην λογοδοσία για να υπάρξουν διώξεις στο μέλλον και να στείλουμε ένα μήνυμα στις βορειοκορεατικές αρχές πως τα εγκλήματα αυτά δεν θα γίνονται πλέον ανεκτά. Αυτό συνέβη και μετά την ε, εποχή της ναζιστικής Γερμανίας όταν είχαν ξεκινήσει σχέδια διώξεων και το γνώριζαν αυτό ήδη οι ηγέτες. Οπότε θα πρέπει να σχεδιάσουμε έναν μακροπρόθεσμο οδικό χάρτη για την δίωξη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και να αντιληφθούμε ρητός ποιες είναι οι καλύτερες επιλογές για το ποιο είναι το επίπεδο ευθύνης και εγκλημάτων που αναζητούμε και ποιες περιόδους καλύπτουν. Αυτό πρέπει να γίνει ε, για να μην είμαστε και απροετοίμαστοι σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος και πιθανής ε, επανένωσης. Γνωρίζουμε πως ε, και η Νότια Κορέα έχει υπογράψει την, το καταστατικό αυτό της Ρώμης, αλλά βεβαίως παρά το ότι υπάρχουν σχέδια για επανένωση, αυτά δεν περιλαμβάνουν κάποια απόδοση δικαιοσύνης για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Πρόκειται για κάτι το καινούριο, το οποίο πρέπει βεβαίως να δούμε και η κοινωνία των πολιτών έχει δείξει πως ε, μπορούμε να έχουμε κάποιες νέες προσεγγίσεις και η διεθνής κοινότητα πρέπει να φροντίσει η διαδικασία αυτή η λογοδοσίας να μην επισκιαστεί από πολιτικούς συμβιβασμούς που πιθανώς προκύψουν στο πλαίσιο της ε, ενοποίησης. Οπότε χρειάζεται ένα σχέδιο το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τον ρόλο της ε, Νοτιοκορέας, ε, της διεθνούς κοινότητας, το γεγονός πως υπάρχουν και αλλοδαποί μεταξύ των θυμάτων της Βόρειας Κορέας και βεβαίως οι παραβιάσεις, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, έχουν ξεκινήσει τη δεκαετία του 1950. Το ζήτημα αυτό το χρονικό τώρα με φέρνει στο επόμενο θέμα που αφορά ακριβώς ε, την δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην περίπτωση που υπάρξει παραπομπή εκεί πέρα. Η Εξεταστική Επιτροπή, όπως είπαμε, αναφέρθηκε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, δεν μπορούμε όμως να αγνοούμε τις προκλήσεις μιας τέτοιας παραπομπής. Όπως ε, είπαμε, αυτό είναι δυνατόν μόνο μέσω μιας παραπομπής μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας και όλοι γνωρίζουμε ποιες είναι οι χώρες που ασκούν βέτο εκεί πέρα και ποιες είναι οι πολιτικές προκλήσεις. Όμως, ακόμα και στο καλύτερο σενάριο που θα συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να λάβουμε υπόψη το θέμα των ε, χρονικών περιορισμών. Δηλαδή, είναι υποσυζήτηση το εάν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα μπορεί να εξετάσει εγκλήματα που διαπράξαν πριν από τον Ιούλιο του 2002. Είναι μεγάλο ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε. Στην περίπτωση επανένωσης, ε, μια που η Νότια Κορέα έχει κυρώσει, όπως είπαμε, τις συμφωνίες της ε, Ρώμης, είναι και πάλι συζητήσιμο το εάν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα μπορεί να εξετάσει εγκλήματα που διαπράχθησαν πριν από την ε, ενοποίηση. Γιατί, όπως είπαμε, ξεκίνησαν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από δεκαετία του 1950 και έτσι θα μείνουν πολλές δεκαετίες εκτός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να εξακριβώσουμε το εάν θα μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη μόνη της η Νότια Κορέα ενώ θα έχει και την ε, πίεση την οικονομική και των ζητημάτων ασφαλείας της επανενοποίησης ή αν θα χρειαστεί τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Επίσης, η Εξεταστική Επιτροπή ε, πρότεινε την ε, σύσταση ενός ειδικού δικαστηρίου μέσω του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης που θα βασίζεται στην αρχή της καθολικής δικαιοδοσίας και του ψηφίσματος ε, ενωμένη για την ειρήνη που ηρωνικά βεβαίως είχε συνταχθεί επί πολέμου της ε, Κορέας. Βεβαίως ε, αναγνωρίζουμε πως είναι μικρές οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο γιατί βεβαίως θα δημιουργούσε ένα προηγούμενο για άλλες χώρες αλλά ακόμα και στο καλύτερο σενάριο που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο υπάρχει η ανάγκη της ε, στήριξης ε, της ε, χώρας που είναι μάλλον απίθανο να συμβεί από τη Βόρεια Κορέα. Μία άλλη επιλογή θα ήταν να αρχίσουμε να εξετάζουμε συγκεκριμένα εγκλήματα όπως οι απαγωγές. Πρέπει να θυμόμαστε πως οι περισσότερες από τις απαγωγές έγιναν σε νότιο-κορεατικό και ιαπωνικό έδαφος από βορειοκορεάτες πράκτορες. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα οι δύο αυτές χώρες να ξεκινήσουν κάποιες έρευνες για αυτά τα εγκλήματα, όμως δεν το έχουν κάνει ακόμα. Οπότε είναι κάτι, είναι μια επιλογή η οποία θα πρέπει να συζητηθεί. Θα είναι κάποια παραδείγματα λοιπόν των επιλογών που υπάρχουν στα διεθνή φόρα. Οι προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών Κοιτάξτε, έχουν δείξει πως ε, κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν. Η Εξεταστική Επιτροπή δεν υπήρχε το 2012, ξαφνικά όμως ε, συναισθάθη. Οπότε υπάρχει η δυνατότητα λογοδοσίας, δεν υπάρχει μόνο ο ΙΕ, υπάρχουν ε, διαφορετικοί μηχανισμοί που θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε. Όλα αυτά θα συζητηθούν ε, από την ε, ομάδα ανεξαρτήτων ειδικών του ΟΗΕ και οπωσδήποτε θα είμαστε σε στενή επαφή μαζί τους όπως ε, έκανε η κοινωνία των πολιτών και πριν με την ε, Εξεταστική Επιτροπή. Έτσι θα περάσουμε στο επόμενο επίπεδο της συζήτησης για τη λογοδοσία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κατερίνη. Ακολουθεί ο προσκεκλημένος μας από την Νότια Κορέα ο κύριος Λί Ιούγκ Χουν πρέσβης για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη Δημοκρατία της Κορέας να υπενθυμίσω τη μοναδική θέση και τον ρόλο της ε, Νότιας Κορέας Ζητήσαμε και από την Αντιπρόεδρο την κυρία Μόγκερίνη να χρησιμοποιήσει την δυνατότητα, τις δυνατότητες της Νότιας Κορέας για να διαμορφώσει την στρατηγική μας για τη Βόρεια Κορέα. Ο Δ. Λί ορίστηκε πρέσβης ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ε, Νότιου Κορέας το 2015. Πριν από αυτό είχε πανεπιστημιακή σταδιοδρομία και ήταν και συμπρόεδρος μιας ε, ομάδας που λεγόταν «Σώστε την Βόρεια Κορέα» και προστάτευε πρόσφυγες από την Βόρεια Κορέα. Μπορεί έτσι λοιπόν να μας ε, δώσει την δική του άποψη για την κυβέρνηση της ε, Βόρειας Κορέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μεγάλο ταξίδι που έκανε για να μας μιλήσει σήμερα. Έχετε τον λόγο κύριε Λύη. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ επίσης και τα μέλη ε, καθώς επίσης και τη Γραμματεία που οργάνωσαν αυτό το πολύ σημαντικό εργαστήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα καθώς επίσης και δεύτερον για την πρόσκληση Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τα συλληπιτήριά μου για τα θύματα του πρόσφατου τρομοκρατικού χτυπήματος εδώ στις Βρυξέλλες. Ε, η Κορέα θρυνεί για τα θύματα και ε, τους ε, συγγενείς τους και χαιρετίζουμε την κυβέρνηση του Βελγίου αλλά και το λαό της ε, για το θάρρος ε, που επέδειξαν σε αυτές τις σίγουρα πολύ δύσκολες εποχές. Δεν υπάρχει θέση για τέτοιες πράξεις βαρβαρότητας. Είναι σίγουρα μια πράξη δηλίας και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεριζώσουμε μια, ε, μια για πάντα από το πρόσωπο της γης. Ταυτόχρονα όμως μπορούμε να πούμε το ίδιο και για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ε, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οπουδήποτε στον πλανήτη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να ξεριζώσουμε με κάθε τρόπο. Το 1945 όταν τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είμαι σίγουρος ότι πολλοί άνθρωποι είχαν, οι άνθρωποι είχαν σοκαριστεί ε, βλέποντας τα όσα είχαν γίνει σε μέρη όπως είναι το Auschwitz αλλά και σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο βαθμός ε, της κατάφορης παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν απαράδεκτος και αυτό φάνηκε στη συνέχεια με τη δίκη της Νιρεμβέργης καθώς επίσης και το 48 με την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αντικατοπτρίζει λοιπόν το αίσθημα των ανθρώπων που οδήγησε σε αυτές τις εξελίξεις και στη συνέχεια στα υπερχόμενα χρόνια υπήρχαν πάρα πολλές συμφάσεις και νομοθεσίες που υιοθετήθηκαν ώστε να αντιμετωπιστούν οι συγκεκριμένες ε, προκλήσεις των σοβαρότερων απειλών προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια όπως είναι για παράδειγμα το Apartheid ε, στην Νότιο Αφρική, η γενοκτονία στη Ρουάντα, οι, Χμερ, οι Ρούς ε, ε, στην Καμπότζη, Ένα μέρος το οποίο μπόρεσε να ξεφύγει όμως από αυτές τις διεθνείς προσπάθειες για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν η Βόρεια Κορέα παρόλο που κάποια ε, από τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί εκεί θεωρούνται από τη διεθνή κοινότητα όσο τα χειρότερα. Πώς κάτι τέτοιο έχει επιτραπεί. Για ποιο λόγο η Βόρεια Κορέα καταφέρει να ξεφεύγει ε, της προσοχής. Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν συναυλίες των YouTube ε, για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για ποιο λόγο άνθρωποι όπως ο George Clooney, η Αντζελίνα Ζολή δεν μιλούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα. Ακριβώς επειδή η Βόρεια Κορέα θα μπορούσαμε να πούμε είναι η πιο κλειστή κοινωνία του πλανήτη. Κανένας δεν μπορεί να βγει, κανένας δεν μπορεί να μπει. Αυτοί οι οποίοι βγαίνουν είναι φυσικά οι θαραλέοι αποστάτες που πηγαίνουν προς την Κίνα και αυτό είναι μια άλλη ιστορία σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί αρχικά στην προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα και κατά δεύτερον η ζωή που πρέπει να υπομείνουν στην Κίνα διότι θα ξέρετε ότι πάνω από το 70% των αποστατών είναι γυναίκες και ένα μεγάλος αριθμός εξ αυτών υπόκεινται σεξουαλική βία μεταξύ αυτών και βιασμούς. Με την Βόρεια Κορέα δεν έχουμε εικόνες και γι' αυτό το λόγο μπορεί και ξεφεύγει η χώρα άλλες ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για αυτές έχουμε φωτογραφίες, έχουμε βίντεο, όμως στην περίπτωση, στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας έχουμε μονάχα τις μαρτυρίες ε, ανθρώπων, δεν έχουμε εικόνες, αλλά επειδή δεν μπορούμε να το δούμε και μονάχα το ακούμε από τις φωνές των θυμάτων, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πραγματοποιείται κάτι τέτοιο. Λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή που έχουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση. για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Η πυρηνική δοκιμή αλλά και το πυρηνικό πρόγραμμα και η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αλληλένδετα. Πολύ απλά είναι δύο σημαντικά εργαλεία για το καθεστώς της Βόρειας Κορέα ώστε να μπορέσει να αυτοδιατηρηθεί, για να μπορέσει να επιβιώσει τα πυρηνικά όπλα είναι για εξωτερική χρήση, ενώ για εσωτερική χρήση είναι η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Βόρεια Κορέα δεν είναι ανόητη. Έχουν δει τι συμβαίνει, τι παθαίνουν οι δικτάτορες που δεν έχουν ε, πυρηνικά όπλα. Ο Σαντάμ Χουσέιν, για παράδειγμα. Ο Μωαμάρ Γκαντάφη. Πέφτουν. Έτσι λοιπόν είναι αποφασισμένοι να έχουν πυρηνικά όπλα, διότι με τα πυρηνικά όπλα οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας πιστεύουν ότι κανείς δεν μπορεί να τους αγγίξει και θα μπορέσουν να συνεχίσουν με ε, τις επερχόμενες γενιές της δυναστείας των Κιμ. 20-30 χρόνια ακόμα αυτής της ε, δυναστείας και θα κλείνουμε έναν αιώνα δυναστείας των Κιμ. Ήδη κλείνουμε 70 χρόνια. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι για εσωτερικό σκοπό, ούτω ώστε να είναι σίγουροι ότι δεν θα έχουν προκλήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο το καθεστώς. Δεν ενδιαφέρονται για την οικονομική ανάπτυξη και για το καλό του λαού. Αν τους ένοιαζε, θα το είχαν κάνει εδώ και καιρό. Ίσως να σας σοκάρει μερικούς που δεν το γνωρίζετε, όμως η οικονομία της ε, Βορείου Κορέα ε, με βάση το ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερη σε σχέση ε, της Νότιας Κορέας μέχρι το 1974. Και σκεφτείτε πού είναι τώρα η κατάσταση των δύο οικονομιών. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες όπου η ε, διεθνής ε, κοινότητα έτεινε ε, χείρα βοηθείας προς την Βόρεια Κορέα. Όμως η Βόρεια Κορέα δεν ανταποκρίθηκε διότι δεν ενδιαφέρεται, διότι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης απειλούν το καθεστώς. Για να διατηρήσει λοιπόν το λαό υπό έλεγχο, ούτως ώστε να μην γύρει προκλήσεις, καταφεύγει στις πιο κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε δει ποτέ. Τα Ηνωμένα Έθνη, όπως δηλώθηκε και προηγουμένως, έχουν υιοθετήσει και ιδιαίτερο στο Συμβούλιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποφάσεις από το 2003, το 2004 υπάρχει ο ειδικό απεσταλμένος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στη Βόρεια Κορέα. Έχουμε την απόφαση του 2005 και από τότε που εκδόθηκε η έκθεση ε, της ε, Εξεταστικής Επιτροπής και αυτό υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο ΙΕ λοιπόν είναι ιδιαίτερα ενεργός για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου. Η έκθεση λοιπόν επέφερε μια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα και με τον τρόπο με τον οποίο η διεθνής κοινότητα με βάση τον ΟΗΕ αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θεωρώ ότι όλο αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Ναι, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα βιωσιμότητας των κυρώσεων και το πώς θα, κατά πώς θα, λειτουργήσουν στη Βόρεια Κορέα. Υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Πιέζουμε τη Βόρεια Κορέα ε, στον τοίχο. Θα πρέπει να επιβραδύνουμε λιγάκι, να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με τη Βόρεια Κορέα. Το κάνουμε αυτό για δεκαετίες όμως δεν απέφερε αποτελέσματα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να επικεντρωθούμε στη λογοδοσία, να συνεχίσουμε την πίεση προς τη Βόρεια Κορέα, γιατί διότι για πρώτη φορά η Βόρεια Κορέα δείχνει ότι δεν είναι σε βολική κατάσταση. Η το ήρξαν αρκετές του Συμβουλίου ασφαλεία κυρώσει ε, πέντε ω τώρα ε, για τι ε, πυρηνικέ δοκιμές τη χώρας, όμω, δεν υπήρχε καμία ανταπόκριση. Η Βόρεια Κορέα παραμένει σκληρή στη στάση τη Όταν όμως το ζήτημα αφορά την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οποιαδήποτε αναφορά για παραμπο, του ζητήματος ε, μεταξύ και του Κιμ ε, Un στο ποινικό δικαστήριο, στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τότε ανταποκρίνεται. Και για οποιονδήποτε λόγο αυτό φαίνεται πως λειτουργεί. Και για αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε μια στοχευμένη προσπάθεια για να αυξήσουμε την πίεση. Αν θυμάστε καλά, ε, με το Apartheid στην Νότια Αφρική το 1994 δεν καταργήθηκε απλά ε, το Απαρτχάιτ και ο ε, Νέρσον Μαντέλα κατάφερε να επανεκλεγεί. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια διεθνής, διεθνούς πίεσης. Θυμάμαι πανεπιστημίου πόλη στη δεκαετία του 90 να ασκούν ε, πίεση σε εταιρείε όπως είναι για παράδειγμα η Νεστλέ για να μην κάνουν επενδύσεις στη Νότια Αφρική ομάδες κρίκετ, ράγμπι δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διεθνείς αγώνες. Δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει στην περίπτωση της Βόρειας Κορέας. Η Βόρεια Κορέα συνεχίζει ε, να συμμετέχει σε διεθνείς ε, αγωνιστικές ε, εκδηλώσεις η κυρία Κατερίνη και η δόκτωρ Μπέκοβα ανέφεραν μερικά βήματα τα οποία θα μπορούσαμε ε, να κάνουμε στο πλαίσιο της λογοδοσίας. Ναι, σίγουρα το καλύτερο βήμα θα ήταν ε, το ε, Συμβούλιο Ασφαλείας να παραπέμψει την υπόθεση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όμως εξαιτίας της Κίνας αλλά και της Ρωσίας ε, και του δικαιώματος αρνησικηρίας, κάτι τέτοιο δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό στο εγγύς μέλλον. Όμως θα ήθελα να προσθέσω στην περίπτωση της Κίνας ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε εκεί είναι ότι πρόκειται για μια χώρα που θέλει να ανταγωνιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ε, μια υπερδύναμη. Θέλει να έχει ε, ένα ρόλο παγκόσμιας ηγεσία και το ε, με την παραπομπή της υπόθεσης του Νταρφούρ αλλά και το 2011 με τη Λιβύη ε, η Κίνα ε, συμφώνησε με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο όμως έτσι δεν μπορούμε να λούμε ότι δεν θα συμβεί ποτέ συμφώνησε στη Λιβύη και στο Νταρφούρ οπότε αν αλλάξουν οι συνθήκες ακολουθήσει μια πέμπτη, έκτη πυρηνική δοκιμή τότε δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν θα διατηρήσει την τωρινή της τάση η Κίνα. Και άλλωστε αυτό φαίνεται άσχημα στην εικόνα της Κίνας ως ε, ε, παγκόσμιος ηγέτας, ηγέτης. Η Κίνα λοιπόν πρέπει να είναι μια ήρεμη δύναμη. Πρέπει να δείξει ότι αντιπροσωπεύει ορισμένε πανανθρώπινες αξίες όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και γι' αυτό το λόγο ελπίζω ότι κάποια στιγμή η Κίνα θα κάνει στροφή 180 μοιρών και θα υιοθετήσει αυτό το ζήτημα ως κάτι το οποίο θα πρέπει η Κίνα να ξεπεράσει για να γίνει πραγματικός ηγέτης και ευελπιστώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει την προσπάθειά της για να πείσει την Κίνα ούτω ώστε να βρίσκεται, να βρίσκεται στη σωστή πλευρά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα. Αναφέρθηκε επίσης πριν ότι μπορούν να γίνουν παραπομπές για χώρες ε, που ε, είναι μέλη του καταστατικού της Ρώμης σε περίπτωση που υπάρξουν παραβιάσεις ε, πολιτών της Βόρειας Κορέας. Η Βόρεια Κορέα δεν, έχει, ε, δεν είναι μέλος του καταστατικού της Ρώμης, όμως γνωρίζουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρες όπου υπάρχουν ε, εργάτες από τη Βόρεια Κορέα και το ερώτημα είναι εργάζονται υπό τις ίδιες συνθήκες με τις οποίες εργάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Σίγουρα όχι. εφαρμόζεται ο νόμος εξίσου. Ε, ε, είστε από την Πολωνία. Συγγνώμη, από την Πολωνία. Στην Πολωνία λοιπόν έχουμε εκατοντάδες βορειοκορεάτες εργάτες, στην Μάλτα επίσης. Και ίσως το ζήτημα αυτό να επεκτείνεται. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Μάλτας κινέζικο εργαστήριο ενδυμασίας απασχολεί βορειοκορεάτες εργαζόμενους. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει προσεκτικά για να διασφαλίσει ότι το εργατικό δίκαιο δεν παραβιάζεται και σε περίπτωση που συμβαίνει ιδιαίτερο σε χώρες που έχουν ε, εγκρίνει το καταστατικό της Ρώμης, τότε θα πρέπει το ζήτημα αυτό να παραπευθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και επίσης το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο από μόνο του με άδεια θα μπορούσε να ξεκινήσει έρευνα το παραπομπή του Συμβουλίου Ασφαλείας από την πλευρά του Συμβουλίου Ασφαλείας ίσως να μην είναι η μόνη εναλλακτική για να στραφούμε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες που αναφέρθηκαν όσον αφορά ε, την ε, ε, σύσταση δικαστηρίου από την Γενική Συνέλευση και αυτό είναι εφικτό στο πλαίσιο του καταστατικού διότι σε περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν λάβει δράση σε μια κατάσταση που ίσως αποτελεί απειλή για τη διεθνή ειρήνη και νομίζω ότι η παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα αποτελεί απειλή τότε πιστεύω ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να στραφεί στην απόφαση ε, United for Peace και να ε, δημιουργήσει ένα δικαστήριο για το θέμα αυτό. Η διεθνής δικαιοδοσία είναι ένα άλλο θέμα. Σίγουρα δεν είναι σύνηθες οι χώρες να ε, στρέφονται σε αυτό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το Ισπανικό Δικαστήριο το οποίο ε, δίκασε τον ε, Πινοσέτ και νομίζω ότι και βελγικά δικαστήρια προσπάθησαν να δικάσουν Χούτου από την ε, Ρουάντα λόγω της γενοκτονίας και αυτή λοιπόν είναι μια ακόμα εναλλακτική όσον αφορά τη λογοδοσία και την εφαρμογή των κυρώσεων. Δεν θα συζητήσω για άλλους ε, μηχανισμούς, όμως υπάρχουν που μπορούν να πιέσουν ε, την ε, Βόρεια Κορέα. Δεν έχει λοιπόν έρθει η ώρα να μην συζητούμε σχετικά με το αν λαμβάνουν χώρα παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να συλλέξουμε κι άλλες πληροφορίες γι' αυτό. Υπάρχουν εκατοντάδε υποθέσεις από καταθέσεις διασωθέντων. Δεν είναι ώρα να συζητήσουμε σχετικά με το αν αυτό συμβαίνει ή όχι. Έχουμε αρκετές αποδείξεις. Έχει έρθει λοιπόν η ώρα να μιλήσουμε σχετικά με το τι θα κάνουμε για αυτό ποια είναι τα μέτρα λογοδοσίας, ποια είναι τα ε, μέτρα πίεσης. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε άλλα 5-10 χρόνια. Αν το πούμε αυτό στους ανθρώπους, ε, τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα στρατόπεδα της ε, Κορέας που αγωνίζονται κάθε μέρα να επιβιώσουν ε, και να τους πούμε ότι σε 5-10 χρόνια η κατάσταση ίσως να βελτιωθεί. Δεν νομίζω ότι ότι ε, θα χαρούν ε, για αυτή την είδηση. Η υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη Βόρεια Κορέα αποτελεί δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την Κορέα, για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει ένα σκληρό αγώνα εναντίον αυτών των υποθέσεων και το πώς θα αντιμετωπίσουμε την υπόθεση της Βόρειας Κορέας είναι μια δοκιμασία σχετικά πάνω στα όσα έχουμε δημιουργήσει και θα πρέπει να συνεχιστεί και στον 21ο αιώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καθηγητά Λί. για την πολύ ζωντανή σας παρουσίαση όσον αφορά τα, ε, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ε, πρόκληση της επιδίωξης λογοδοσίας ε, και τέλος ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τζούλιαν Βίλσον που είναι επικεφαλής του τμήματος για την Ιαπωνία, την Κορέα, την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία ε, από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, θα μας παρουσιάσει τις ευρωπαϊκές προσπάθειες ώστε να ε, υπάρξει λογοδοσία στη ΟΝΟΙΕ, τις προκλήσεις ποια είναι η ε, πολιτική μας και ποιες είναι οι προβλέψεις για το μέλλον. Έχετε το λόγο κύριε Βίλσον. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Μεγάλη μου χαρά που έχω την ευκαιρία να σε απευθύνω το λόγο και να συναντήσω και τον πρέσβη της Νότιας Κορέας για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε αυτό το δύσκολο θέμα. Εμείς, ο Πρόεδρος ε, ανέφερε στην εισήγησή του ποιος είναι ο ρόλος μας απέναντι στη Βόρεια Κορέα. Να σας δώσω μια γενική εικόνα. Ο στόχος είναι να έχουμε δραστήριο και επικοδομητικό ρόλο όπως αυτό που είπε ο Πρόεδρος, και αυτό βασίζεται στην... βασίζεται μάλλον στην σε κίνητρα και αντικίνητρα ανάλογα με τις αντιδράσεις της Βόρειας Κορέας. Το ψήφισμα του ΟΗΕ δείχνει αυξανόμενο ενωμένο διεθνέ μέτωπο, ε, το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Είναι μια ευκαιρία για να ασκήσουμε πιο μεγάλη πίεση στην Βόρεια Κορέα απέναντι σε αυτή την κρίσιμη και πιεστική θέση θα πρέπει να πούμε ότι το, η Βόρεια Κορέα κατανοεί πάρα πολύ καλά ότι η θετική συνεργασία είναι δυνατή αν οι ενεργές της εγγυηθούν κάτι τέτοιο και αν το κλίμα βοηθά. Πρέπει να σας πω ότι επί του παρόντος δεν ίσχυε κάτι τέτοιο Πρόεδρε. Η στήριξη εκτός ε, συνεχίζεται ε, για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά ε, θέλουμε, παίζουμε και ηγετικό ρόλο, ε, ρόλο ε, όσον αφορά τα θέματα που εξετάσατε όλο το πρωινό σήμερα, ε, το πυρηνικό πλωστάσιο, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχουν ε, ε, ετήσιες εκθέσεις ε, και αυτό που είναι ενδιαφέρον όσον αφορά το συνασπισμό για ένα ενωμένο μέτωπο κατά της Βόρειας Κορέας είναι ότι κάθε ε, είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά όλο είναι και περισσότεροι υπεψηφίζουν τα ψηφίσματα αυτά στην Γενέβη και αυτό στέλνει ένα μήνυμα με μια έκκληση για δράση και γι' αυτό είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανοιχτή, όπω σχολίασαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ. Έχει οριστεί ο κύριο Δέρα μα ο ειδικός εισηγητής και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία ε, που έχουμε τα τελευταία έξι χρόνια συμπεριλαμβανομένη εργασία του στη διάρκεια και μετά την Επιτροπή έρευνα, Αλλά έκτοτε δεν έχουμε λάβει πληροφορίε που μα λένε ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει βελτιωθεί. Ε, Σοβαρέ παραβιάσει συνεχίζονται και πρέπει λοιπόν να διατηρηθεί η πίεση όχι μόνο στον τομέα της ε, ετήσιας έκθεσης μέσω του ΟΙΕ αλλά και μέσω της πίεσης του ΟΙΕ για συνέχιση του διαλόγου καθώς και με, υπό την απειλή της παραπομπής στο Διεθνές ε, Δικαστήριο της Χάγης. Ε, πρέπει να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος. Έγινε πολιτικός διάλογος πέρυσι, Πρόεδρε, όπου μάλιστα συζητήσαμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θέμα προτεραιότητας μαζί με τις πολιτικές ε, για τις, ε, τα πυρηνικά όπλα της χώρας. Όμως φέτος δεν θα γίνει τέτοιος διάλογος και επίσης μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι δεν θα γίνει ούτε και διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, φέτος για προφανείς λόγους. Ε, στην τελευταία συνεδρίαση προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στην έκθεση του ειδικού απεσταλμένου, αλλά δεν τα καταφέρουμε. Ωστόσο, καταγγέλουμε τις καταχρήσεις, καταγγέλουμε τα όσα συμβαίνουν εκεί και εστιάζουμε στη βελτίωση των σχέσεων. Προσπαθούμε να βρούμε κάποια κοινή ατζέντα για συνεργασία πριν από τις πυρηνικές δοκιμές, το προσπαθήσαμε αυτό, όπου αναζητούσαμε δυνατότητες για συνεργασία και ε, είχαμε πάνω από 100 συστάσεις στην ε, ετήσια περιοδική μας ε, έκθεση του 2014. Επιμένουμε για τεχνική βοήθεια εάν οι όροι και προϋποθέσεις και οι εταίροι μας δείξουν ειλικρινή πρόθεση να βελτιώσουν την κατάσταση στη χώρα. Φοβούμαι πως αυτό δεν συμβαίνει τώρα, άρα δεν έχουμε κανένα σχέδιο για αυξημένη συνεργασία επί του παρόντος. Ακόμα και αν συντονίζουμε τις κυρώσεις και τις ποινές, προσπαθούμε να αποφύγουμε να πλήξουμε το ευρύ κοινό και αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει η ανθρωπιστική βοήθεια όταν χρειάζεται. Το ίδιο ζήτησε και η Επιτροπή Έρευνας. Φέτος δεν έχουμε μεγάλη αισιοδοξία. Ε, γιατί συνεχίζονται οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζονται οι πυρηνικές δοκιμές ε, και οι εκτοξεύσεις ε, πυράβλων. Αλλά φαίνεται ότι είμαστε πιο ομόφωνοι να πιέσουμε τη χώρα αυτή να ακολουθήσει διαφορετική πορεία. Ίσως αυτό να είναι ένα στοιχείο, μια ευκαιρία, ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στα όσα ζητάμε. Ε, και στα επιχειρήματά μας. Θέλω να υπογραμμίσω και τη στήριξη τη Κίνα στο τελευταίο πακέτο κυρώσεων που ήταν ε, εστιασμένο στα πυρηνικά και είναι μια ευκαιρία για να συνεργαστούμε με την Κίνα για όλες τις πτυχέ πολιτική στη Βόρεια Κορέα και αυτές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο προηγούμενο ομιλητή είπε ότι θα βρούμε ότι υπάρχουν, υπάρχει μέχρι βαθμό συμφωνίας και η Κίνα θα παίξει σημαντικό ρόλο σε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη χώρα αυτή. Οτιδήποτε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε για να συνεργαστούμε με την Κίνα και να συγκλίνουν οι πολιτικές μας απέναντι στη Βόρεια Κορέα θα είναι κάτι το οποίο θα επικροτήσουμε. Τέλος όμως θέλω να επιστήσω την προσοχή σας ότι πρέπει να τονίσουμε τις πιέσεις και τις κυρώσεις έτσι ώστε η Βόρεια Κορέα να έχει μια σταθερή και ισχυρή ε, ένα ισχυρό μήνυμα το αδιαφυσβήτητο από όλα τα μέρη ότι πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις και να πάψει τις πολιτικές που οδηγούν σε εγκλήματα ε, και σε βίες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να σχολιάσω δε, το θέμα των εργαζομένων της Βόρειας Κορέας στην Ευρώπη, γιατί αναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές. Αυτό το θέμα έχει προκύψει εντόνως φέτος ε, έχουμε συζητήσει με τα κρατημέλη, δεν μπορώ να σας δώσω τώρα άμεσα συγκεκριμένες λεπτομέρειες, γιατί πρόκειται για εμπιστευτικές συζητήσεις για τα κρατημέλη, όμως εργάζονται για αυτό το θέμα, το οποίο εμπίπτει στη δική τους εντολή, στις δικές τους αρμοδιότητες. Η Ένωση δεν μπορεί να κάνει κάτι για τις θεωρήσεις κτλ. Οπότε κάπως περιορισμένες πληροφορίες μπορώ να σε μοιραστώ μαζί σε αυτή τη στιγμή. Όμως αυτό που διαπιστώσαμε σαφές είναι ότι ο αριθμός... Ε, οι αριθμοί των εργαζομένων είναι αρκετοί, αν και όχι τόσο μεγάλοι όσο στην Κίνα ή στη Ρωσία, και ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να αντιμετωπίσουν το θέμα. Είναι περιορισμένο ο αριθμό των Βορειοκορεατών εδώ, αλλά ε, τα κράτη-μέλη θέλουν να το αντιμετωπίσουν το θέμα ε, για να μην γίνει μεγαλύτερο. Ο προηγούμενο ομιλητή είπε ότι ίσω αν, δεν δράση, ίσω να αναπτυχθεί υπερβολικά Μπορώ να σας πω ότι η τάση είναι ε, ναι, να εντοπίσουμε το πρόβλημα είναι μικρότερο από ό,τι σε άλλες χώρες και αναζητώνται λύσεις ε, μεμονωμένα από τα κρατημέλη, ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε καθένα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την επίλυση του προβλήματος και να μην αυξηθεί το πρόβλημα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τζούλιαν. Και τώρα τα μέλη μπορούν να πάρουν το λόγο. Ή άλλοι συμμετέχοντες. Ο πρώτος που θέλει να πάρει το λόγο είναι ο κύριος Κρίστιαν Πρέντα που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι είμαι ικανοποιημένος που διοργανώθηκε η σημερινή ημερίδα ε, μελέτης γιατί ακριβώς πριν ένα χρόνο προσπάθησα να πείσω τους συναδέλφους ότι μέσω του Επισκόπου Γιούνα που είναι γνωστός ε, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των, ανθρωπίνων, ε, Βορειοκορεατών ε, ε, έπρεπε να κληθεί εδώ. Δυστυχώ δεν έπεισε αρκετού συναδέλφου να στηρίξουμε αυτή την υποψηφιότητα για το βραβείο Ζαχάροφ. Είναι κάπω κρίμα γιατί κριτώ την ιστορία του βραβείου Ζαχάροφ που είναι πολύτιμο βραβείο. Ποτέ δεν δώσαμε βραβείο σε κάποιον ο οποίο υπερασπίστηκε τα δικαιώματα των Βορειοκορεατών. Και είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό διότι πρόκειται για έναν απολυταρχισμό εγκληματικού τύπου όπως κάθε πολιταρχισμός. Είναι ένα καθεστώς που βλέπει να αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο ο λοιμός, να επιδεινώνεται είναι ένα είδος ε, ηθελημένης ε, σκλαβιάς, δουλείας, γιατί δεν υπάρχει καμιά αντίσταση στη χώρα, καμιά αντιπολίτευση. Ε, δυστυχώς λοιπόν δεν έγινε δεκτή η πρόταση στις ομάδες μου να στείλουμε μια αποστολή στην Νότια Κορέα ώστε να ενθαρρύνει τους όσους εκεί αγωνίζονται για τις τα δικαιώματα των Βόρειο Κορεατών Φαίνεται να υπάρχει μεγάλη νοσταργία για τον κομμουνισμό, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε αυτό το κοινοβούλιο. Και λυπούμε που δεν είναι εδώ κανένα κομμουνιστή σήμερα για να μα εξηγήσει πώ ε, βλέπει, ποια είναι η γνώμη του για αυτό το τελείω ανεύθυνο κομμουνιστικό καθεστώ, το οποίο ηγείται ένα ηγέτη που ανα πάσα στιγμή κινδυνεύει να ξεκινήσει έναν πόλεμο ακόμα και θέλετε γιατί είναι τόσο τρελός που, και παράλογος που οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και με μια πλήρη ανευθυνότητα από πλευράς, ιδιαίτερα μεγάλη ανευθυνότητα από πλευράς της Κίνας. Και πρέπει να πω ότι η ευθύνη της Κίνας, όπως αναφέρθηκε και με το τελευταίο ψήφισμα που εγκρίναμε τον Ιανουάριο, η ευθύνη της Κίνας είναι πολύ μεγάλη σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε οριακά να πούμε ότι οι Βορειοκορεάτες αισθάνονται θύμα τα του καθεστώτος της Κίνας, όπως και οι Κινέζοι είναι οι ίδιοι θύματα αυτού του άλλου απολυταρχισμού που έχει γίνει πολύ εμπορικός και πολύ αγαπητός στην Ευρώπη ακριβώς για εμπορικούς λόγους. Αυτή είναι η μεγάλη ε, η διαφορά είναι, είναι το καθεστώς ε, του Πεκίνου το οποίο θυσιάζει και τους Βορειοκορεάτες. Εάν οι Κινέζοι συμφωνούσαν να εγκαταλείψουν ε, την σημερινή βορειοκορεατική δυναστεία, τότε η τύχη των βορειοκορεατών θα ήταν ε, τελείως διαφορετική από τη μια μέρα στην άλλη. Αυτό είναι σαφές. Η ευθύνη της Κίνας είναι τεράστια και πρέπει αυτό σαφώς να το πούμε στις ε, πολιτικές μας θέσεις, γιατί και πάλι η αμφισημία στις σχέσεις μας με την Κίνα υπάρχει και ελπίζω ότι στη, διάρκεια του ταξιδιού που θα κάνει η, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στην Κίνα θα υπογραμμιστεί αυτό. Η ευθύνη των Κινέζων είναι μεγάλη. Οι, οι Βορειοκορεάτες είναι θύματα της Κίνας. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρέντα. Επόμενος που θα πάρει το λόγο είναι ο κύριος Ντεμασμάκερ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαστήριο. Βεβαίω δεν χρειάζεται να πείσουμε εαυτούς ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Κορέα. Γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση και το τι γίνεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα στην κομμουνιστική αυτή δικτατορία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πράγματι πως είναι μία από τις πιο κλειστές χώρες αυτού του πλανήτη και δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ασκήσει κάποια σοβαρή επιρροή στο καθεστώς. Είναι πάρα πολύ κλειστό μέρος και έχουμε λίγες άμεσες πληροφορίες. Στηριζόμαστε σε διηγήσεις. Ε, ε, εδώ πέρα η βελγική τηλεόραση έχει ένα πρόγραμμα ταξιδιωτικό. Ε, ο Βάς ταξιδεύει, ο Βάς είναι ο παρουσιαστής, ο οποίος ε, έχει πάει σε διάφορες χώρες στις οποίες δεν μπορούν να πάνε οι απλοί τουρίστες και μία από αυτές ήταν η Βόρεια Κορέα. Τρία χρόνια προσπαθούσε να πάρει άδειε, βίζες κτλ. Και είδαμε την εκπομπή. Μας δείχνει μια χώρα τελείως κλειστή. Και είναι βεβαίω συνεχώ εκεί πέρα υπό την συνοδεία των ανθρώπων του καθιστότος. δεν μπορούσε να μιλήσει απευθεία σε απλούς Νοτιοκορεάτε. Έβλεπε ε, μόνο αυτό το οποίο ήθελε η Νότια Κορέα να δει και πήγε με 100 ερωτήσεις και επέστρεψε με 1000 ερωτήσεις. Είναι λοιπόν μία από τις πιο κλειστές χώρες του πλανήτη. Έχω τώρα κάποιες ερωτήσεις. Αντιλαμβάνομαι πως η Βόρεια Κορέα μέχρι τις αρχές Μαρτίου συνεργαζόταν με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τώρα δεν συμβαίνει αυτό. Ποια είναι η διαφορά στην πράξη λοιπόν μεταξύ της προηγούμενης περίοδου και, και του τώρα. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συμφώνησε ομόφωνα σε νέες κυρώσεις κατά της ε, Βόρειου Κορέας. Ε, Διάσα, μάλιστα πως είναι οι σκληρότερες κυρώσεις εδώ και 20 χρόνια. Τι αντίκτυπο έχουν ε, στον πληθυσμό και στο καθεστώς και, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης ε, τις δικές της ε, κυρώσεις. Ε, το ερώτημα λοιπόν είναι, σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σκεφτεί περαιτέρω και επιπρόσθετες κυρώσεις. Έχουμε επίσης την κατάσταση όπου ακούμε κάποιες, κάποια αισιόδοξα λόγια από πλευρά Κίνας και τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει. Βεβαίω ακούω και άλλα πράγματα, ότι η Κίνα παραδείγματο χάρη ε, ε, στέλνει πίσω τους βορειοκορεάτες πρόσφυγες όσους καταφεύγουν στην Κίνα, εν Γιατί ε, ακούω λοιπόν κάποια αντιφατικά πράγματα, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας διαφωτίσετε εδώ πέρα. Και όσον αφορά τους βορειοκορεάτες εργάτες στο εξωτερικό, μιλήσαμε για ευρωπαϊκές χώρες, αλλά διαβάζω, παραδείγματο χάρη, ότι χιλιάδες Βορειοκορεάτες αυτή τη στιγμή εργάζονται στο Κατάρ όπου χτίζουν ε, τα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2020 σε απάνθρωπες συνθήκες όπου παίρνουν μόνο κλάσμα της αμοιβή του. και κάποιοι το έχουν πει αυτό κρατική σκλαβιά το έχουν περιγράψει. Και βεβαίω εμείς ως διεθνής κοινότητα βλέπουμε να οργανώνεται ένα τσίρκο για το ποδόσφαιρο αλλά πρέπει λίγο να σκεφτούμε ποια είναι η ευθύνη που υπάρχει και τι πληροφορίε έχουμε για αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Σάστρεβίτσος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο Economist ε, πρόσφατα έγραψε ένα ενδιαφέρον άρθρο για την Βόρεια Κορέα. και έκανε κάποιες εκτιμήσεις για το σε ποιο βαθμό είναι λογικές ε, οι αρχές της Βόρειας Κορέας και βασίστηκαν σε κάποιες ε, σχεδιασμένες ε, αντιδράσεις και απαντήσεις της ε, Δύσης και το τι συμβαίνει στην εσωτερική πολιτική της χώρας την οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε κάπως καλύτερα. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ αλλιώς πώς μπορούμε να εξηγήσουμε παραδείγματος χάρη το ότι ακόμα και υπό καθεστώς κυρώσεων ε, εξακολουθεί να επιζεί η οικονομία αυτής της χώρας, ε, έστω σε πολύ κακή κατάσταση και παρακάμπτει τις κυρώσεις μας. Σε ποιο βαθμό λοιπόν Οι κυρώσεις ε, και οι περιορισμοί στο εμπόριο με τη Βόρεια Κορία είναι επιτυχής. Μπορούμε ίσως να έχουμε κάποιες πιο απτές ε, κυρώσεις. για να περιοριστούν κάπως οι αρχές της ε, Βορειοκορέα. Αλλιώ Αλλιώς θα δούμε και την πέμπτη και έκτη και έβδομη πυρηνική δοκιμή. που βεβαίως δεν αφορά την περιφερειακή μόνο κατάσταση, αλλά και την παγκόσμια κατάσταση. Εγώ θα έλεγα πως οι πράξεις αυτές είναι υπολογισμένες και έχουν προβλέψει και μία αντίδραση, ίσως και στρατιωτική από το εξωτερικό. Οπότε το ερώτημά μου είναι, Ποια είναι η αποτελεσματικότητα των ε, κυρώσεων και μήπως ε, θα μπορούσαν να επιβληθούν ακόμη εντονότερες ε, κυρώσεις, βαρύτερες κυρώσεις στη Βόρεια Κορέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να χαιρετήσω κιόλας τον ε, πρέσβη της ε, Δημοκρατίας της Κορέας, τον κύριο Χάν και τους συναδέλφους του. Ήρθε. Εδώ. Α, εδώ ήταν, μάλιστα. Και συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, εγώ θυμάμαι τα τελευταία χρόνια του καθεστώτο Τσαουσέσκου στη Ρουμανία, τέλη τη δεκαετία του 80, όταν έλεγαν ότι ο Τσαουσέσκου προετοίμαζε να φτιάξει πυρηνικά όπλα. Γιατί όλα αυτά τα έχω ξαναζήσει. αυτά τα δικτατορικά συστήματα που οι τα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, πάνε χέρι-χέρι με διάδοση των πυρηνικών όπλων. Συμφωνώ λοιπόν με τον κύριο Πρέζη, τον κύριο Λί, ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο υπομονής και χαίρομαι για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, είναι προσιλωμένη στο να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των αδελφών μας ε, στη Βόρεια Κορέα που υποφέρουν. Πράγματι, όπως είπε και ο κύριος Πρόντα, Πρέντα, πρέπει να δούμε την ευθύνη της Κίνας και της Ρωσίας ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Απαράδεκτη στάση. Δεν είναι δυνατόν να ε, έχουμε την Κίνα κομμουνιστικό καθεστώς ή το πρώην απολυταρχικό καθεστώς ε, της Ρωσίας, την πρώην Σοβιετική Ένωση, να συνεχίζουν την συνενοχή τους. στο απάνθρωπο καθεστώς ε, της ε, Βορειοκορέας. Θεωρώ πως ε, η δημοκρατία της Κορέας, από την άλλη, είναι στρατηγικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πρέπει λοιπόν να αντιταχθούμε πολύ περισσότερο στην Βόρεια Κορέα και να συνεργαστούμε περισσότερο με την Νότια Κορέα. Γιατί μέσω της ε, συνεργασίας και της εμισολάβησης θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάποια αποτελέσματα και να κάνουμε κάποια αποτελεσματικά βήματα κατά των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. κατά του καθεστώτος αυτού του απολυταρχικού, του κομμουνιστικού που μου θυμίζει την κατάσταση της ε, Ανατολικής ε, και της ε, Δυτικής Γερμανίας. Πριν επανενωθούν. Νομίζω και άλλωστε αυτός είναι και ο βασικός στόχος της ε, διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, να δώσω τον λόγο για λίγο μια που οι διερμηνείς μας δίνουν το χρόνο κυρία Μπίρκοβα. Όχι. Όχι, ο κύριος Μπίρς. Α, με χνιδιάσατε. Κύριε Πρόεδρε, πάνω που χαλάρωνα. Τέσσερις ερωτήσεις λοιπόν, στις οποίες θα ήθελα να απαντήσω, αν μου επιτρέπετε. Μία από τις πιο σημαντικές είναι να ρωτήσουμε εάν μπορούν να είναι αποτελεσματικές οι κυρώσεις. Να ξεκινήσουμε εδώ πέρα με το επίπεδο του εμπορίου. 5 δισεκατομμύρια ευρώ με την Κίνα, 34 εκατομμύρια με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε όσο σκληρές και να είναι οι κυρώσεις, δεν στέκει οικονομικά το ότι θα τους κατευθύνουμε με τις κυρώσεις. Αλλά πρέπει παρόλα αυτά να επιμείνουμε γιατί υπάρχει η πολιτική πτυχή και η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το είπαν οι ομιλητές ότι είναι ευαίσθητη σε αυτά η Βόρεια Κορέα. Επίσης τονίζει τη δυνατότητα συνεργασίας με την Κίνα και ξυπακούεται αλλά νομίζω θα πρέπει να το πω όπως είπε και ο πρόεδρος ότι η Νότια Κορέα πάντα ήταν ε, ο βασικός μας στρατηγικός τέρος με εμπόριο 80 δισεκατομμύρια ευρώ ε, εμπορίου ε, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολύ στενές πολιτικές σχέσεις και συνεργαζόμαστε μαζί τους σε καθημερινή βάση. Για το θέμα των εργαζομένων και για την κλίμακα για την ανταλλαγή πληροφοριών. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι εκτιμήσεις, αλλά θα έλεγα πως είναι μεταξύ 50 και 100 χιλιάδων ε, ανθρώπων ε, από την Βόρεια Κορέα που εργάζονται στο εξωτερικό. Ε, τώρα, για ε, εμάς, ε, για τις δικές μας χώρες, θα έλεγα λιγότερο από χίλιους. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να συζητήσουμε το θέμα με τρίτες χώρες για να θίξουμε αυτό το ζήτημα, ε, γιατί αφορά κυρίως άλλες χώρες, αλλά έχουμε και το δικό μας βάρος και θέμα που πρέπει να επιλύσουμε τέλος, κύριε Πρόεδρε οι τακτικές αλλαγές ε, που έγιναν στον διάλογο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ πως είναι ακριβώς ε, τακτικές αυτές οι αλλαγές και όχι ουσιαστικές. Εγώ ήμουν... Ε, είδα αυτή την επίθεση αγάπης θα έλεγα από την Βόρεια Κορέα αλλά δεν είδα κάποια αλλαγή στην ουσία και έχω την αίσθηση πως είναι πολύ σημαντικό για εσάς τους πολιτικούς να μεταφέρεται το μήνυμα ότι δηλαδή το θέμα που μας απασχολεί με τη Βόρεια Κορέα είναι τα όπλα μαζικής καταστροφής, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι το αφήγημα παραμένει αυτό και οποιαδήποτε αλλαγή ε, δεν ε, θα προέλθει όπως είπαμε από αυτό το φύγημα. Και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε και είμαστε τώρα για πρώτη φορά ενωμένοι με την Κίνα και άλλες χώρες και έχουμε μια ευκαιρία να το αλλάξουμε αλλά όπως σας είπα ακόμα είναι μακρύς ο δρόμος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μάλιστα. Ε, να δώσω λόγο τώρα στον κύριο Πρέσβη. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις και το θέμα της Κίνας και το πώς θα πείσουμε την Κίνα. Η Κίνα θεωρεί την Βόρεια Κορέα ως ε, ένα κράτος, ε, μια προστασίας απέναντι στην, ε, στη ΣΥΠΑ. Και Άρα δεν θεωρούν ότι υπάρχει κάποια απειλή από την Βόρεια Κορέα και μία επανένωση της Κορέας θα έχει και τεράστιες επιπτώσεις ε, θετικές ε, στην βορειοανατολική περιφέρεια της Κίνας που έχει μείνει πίσω από την ακτογραμμή. Οπότε αν επανενωθεί η Κορέα και να έχουμε σύνορα εμείς με την Κίνα, με τη Samsung, την LG και τη Hyundai ε, να μπορούν άμεσα να επενδύσουν στην βορειοανατολική Κίνα. Δηλαδή η Κίνα ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά. Οπότε πρέπει να πείσουμε την Κίνα για τα υπέρ της ε, επανένωσης. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω για τις κυρώσεις ε, το εάν ε, πλήττουν περισσότερο την κυβέρνηση ή το λαό. Σε οποιονδήποτε Βόρειο-Κορεάτη ε, μιλήσετε που έχει φύγει από τη χώρα, έχω μιλήσει με πολλούς από αυτούς και όλοι μηδενός εξαιρουμένου θα σας πούν ότι γιατί η Νότια Κορέα δίνει γιατί η διεθνή κοινότητα δίνει τόση βοήθεια στη Βόρεια Κορέα και η Νότια Κορέα. Και ότι αυτά παρατείνουν την ζωή του καθεστώτος και βεβαίως ε, τη, τη δυστυχία του λαού. Αυτό θα σας πούν. Η κατάσταση στο Κατάρ Γύρω στους 200 ε, Βορειοκορεάτες έχουν απελαθεί ήδη, αλλά έρχονται άλλοι. Και όπως είπατε, είναι σημαντικός ο αριθμός αυτών που δουλεύουν σε εργοτάξια. Και αυτές οι απελάσεις, ελπίζουμε, οδηγούν σε βελτίωση των συνθηκών εργασίας ε, όσων έχουν απομείνει ή θα έρθουν από εκεί και πέρα. Αλλά μιλήσατε για μια κρατική σκλαβιά. Κοιτάξτε, ε, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν αλλά δεν πληρώνονται άμεσα. Μπορεί αυτό να γράφει το συμβόλαιο, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει αυτό. Σας ευχαριστώ. Thank you. Uh, yeah, I think uh, one of the points that was raised. Ευχαριστώ. Ένα από τα ζητήματα στο οποίο θα ήθελα να απαντήσω είναι η ευθύνη της Κίνας, η ευθύνη για προστασία. Σε περίπτωση παραπομπής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είπαμε πως αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Κίνα προσφάτως σε σχέση με μια διεθνή θέση για αυτό το θέμα όμως δεν ξεχνάμε και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το ότι μια παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο είναι συζητήσιμο το εάν και κατά πόσον θα συμβεί βεβαίως και πρέπει να αναρωτηθούμε εάν θα εξετάσει τα εγκλήματα πριν από το 2002 ή αν θα ξεκινήσει από εκεί και μετά. Δεν είναι κάτι το δευτερεύον αυτό, είναι μέρος της συζήτησης. Μετά, υπάρχει το θέμα, ναι, η ευθύνη προστασίας, η πρόοδος της Κίνας κτλ, αλλά, όπως υπόθηκε, ακούμε ότι έχουμε περιπτώσεις επαναπροωθήσεων από την Κίνα στη Βόρεια Κορέα και αυτό δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Οπότε εμείς ε, είμαστε εδώ, η διεθνή κοινότητα, τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα. Τελευταίο, όπως είπα, εμείς θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα οδικό χάρτη για αυτά τα εγκλήματα, τις ευθύνε και να δούμε και ως που εκτείνεται χρονικά η δικαιοδοσία οποιοδήποτε τέτοιου μηχανισμού. Σας ευχαριστώ. Κύριος Πάρντο κατόπιν. Δύο παρατηρήσεις να κάνω μόνο. Η μία αφορά την Κίνα. Συμφωνώ με τα όσα είπε ο κύριος Πρέσβης. Πρέπει να εστιάσουμε στην οικονομική ανάπτυξη. Η Κίνα ε, παίζει σημαντικό ρόλο γιατί η Βόρεια Κορέα είναι φτωχή και θα πρέπει να τονιστεί ότι η Κίνα θα ωφεληθεί από την επανένωση. Η Κίνα δεν είναι αντίθετη με την επανένωση, αλλά είναι αντίθετη με την επανένωση και την παραμονή αμερικανικών στατευμάτων ε, στην ε, Νότιο και στη Βόρεια Κορέα. Έχουμε διπλωματικές σχέσεις με την Νότια Κορέα και η Βόρεια Κορέα καθιστά σαφές ότι είναι το τέλος των τις της ειδικής με τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα. Και αυτό καθίσταται σαφές στις βορειοκορεατικές ε, εφημερίδες. Μπορεί να χειραγωγηθεί η επιρροή της Κίνας, ε, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν αποδειχθεί ότι θα έχει ωφέλη η Κίνα αν αλλάξει η κατάσταση. Τώρα, ε, όσον αφορά τις κυρώσεις και αν είναι αυτές επιτυχείς, θα πρέπει να εφαρμοστούν, αλλά η Βόρεια Κορέα θα εξακολουθήσει με τις πυρηνικές δοκιμές, εκτός αν υπάρξει σαφέστερη δέσμευση. Και επανέρχομαι στη δεκαετία του 90 που έχουμε την πρώτη πυρηνική κρίση, συζητήσεις και συνομιλίες με την ε, κυβέρνηση Κλίντον, τεσσεραμερείς κυβερνη... Ε, συνομιλίες ε, μετά εξαμερείς συνομιλίες το 2002, το 2007 συμφωνίες εξαμερείς, το 2009 δεν έχουμε άλλη εμπλοκή, μετά έχουμε και άλλες πυρηνικές δοκιμές Όλο και περισσότερες προκλήσεις λοιπόν θα γίνονται από τη στιγμή που δεν υπάρχουν κυρώσεις. Νομίζω πως ε, θα πρέπει όλα αυτά να προχωρήσουν μαζί. Θα είμαι σύντομη, ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα στην πρώτη μου παρέμβαση. Θα πρέπει να προωθήσουμε για, για ψήφισμα περί και θα ήθελα να αποθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από το, 90, από το 50 μάλλον, δεν υπάρχει συμφωνία και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο. Δεύτερον, για το θέμα της σχέσης ανάμεσα στον, στον ΟΗΕ και την Κορέα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων η στάση της Βόρειας Κορέας για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει αλλάξει, αλλά είναι, ε, εξακολουθεί να είναι άσχημη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δέχεται κάποιους μηχανισμούς όπως ε, η UPR αλλά απορρίπτει άλλο, όπως το, ψηφί, το ψήφισμα που εγκρίνεται κάθε χρόνο ή τον ειδικό εισηγητή για την Βόρεια Κορέα. Είναι μισοανοιχτό ή μισόκλειστο το παράθυρο ανάλογα όπως θέλετε να το δείτε. Σας ευχαριστώ όλα τα μέλη του πάνελ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε την ε, ημερίδα αυτή περί της λυπηρής κατάστασης λέγοντας ότι ο διάλογος ανάμεσα στη Βόρεια Κορέα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ έχει διακοπεί. Πιστεύω ότι ακόμα και για την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να ε, ε, ξαναέρθουμε σε διάλογο με την Βόρεια Κορέα και γι' αυτό ζητάμε την υποστήριξη σας, την υποστήριξη της Νότιας Κορέας, της Δημοκρατίας της Κορέας. Σας ευχαριστώ όλους. Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι.